αποφασίζεται αυτό. Και τροποποιείται έτσι η ημερησία διάταξη. Περνάμε τώρα στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα συμπεράσματα του τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30 Ιανουαρίου 2012. Και χαιρετίζω από αυτού το κύριο Φανρόπαϊ, πρόεδρο της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον κύριο Μπαρόζο, πρόεδρο της Επιτροπής και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο κύριο Φανρόπαϊ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία δύο χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπρεπε να πάρουν δύσκολες και συχνά επώδυνα μέτρα για να σταθεροποιήσουν την Ευρωζώνη. Παρότι αυτό ήταν αναγκαίο και τώρα αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε και να βλέπουμε ότι άξιζε τον κόπο, αναγνωρίζουμε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ικανή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την οικονομική ανάκαμψη. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το Euro Plus. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάρτιο θα εστιάσει στην διαρθρωτική ανάπτυξη. Και οι οικονομίες των περισσότερων χωρών μας αυξάνονται, αναπτύσσονται και αυξήθηκαν μάλιστα και το 2010 και το 2011. Το άτυπο Συμβούλιο μίλησε για την, που έλαβε χώρα μίλησε για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Βασικά εκεί εστιάσαμε τις συζητήσεις. Παράλληλα όμως εγκρίθηκε και το τελικό κείμενο της συνθήκης ESM και μπήκαν τελευταίες πινελιές στη συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και την διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα είδατε από τις δηλώσεις που ενέκριναν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι το ονομάσαμε δημοσιονομική εξυγίανση φιλική προς την ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό το να μειωθεί το χρέο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν οι επενδύσει για το μέλλον. Στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στις πράσινε υποδομέ. Η αύξηση τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μα θα τι κάνει πιο ελκυστικέ και θα μπορέσουν να προσλάβουν ανθρώπου. Η στρατηγική για την ανάπτυξη καλύπτει πολλέ πτυχέ. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι οικονομικέ πολιτικέ και η ανταγωνιστικότητα είναι μια πτυχή, αλλά ειδικέ πολιτικέ οι εθνικέ αρμοδιότητε, από τη μία και οι αρμοδιότητες της Ένωση από την άλλη. Έχουμε τις εξής προτεραιότητες. Πρώτον, το να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση ιδίως για νέου. Την περασμένη εβδομάδα έλαβα μία επιστολή από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ νεότητα όπου μου έγραψαν ότι οι νέοι σε στιγμές κρίσης και οικονομική λιτότητας δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, αλλά επενδύσει. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά κονδύλια για να υπάρξουν σχήματα και προγράμματα μαθητείας και να βοηθήσουμε έτσι τους νέους αλλά και τους νέους επιχειρηματίες. Η ενίσχυση της απασχόλησης είναι κυρίως ευθύνη των επιμέρους χωρών. Αλλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα κάνουμε. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα για την απασχόληση Ω ε, τμήμα του Εθνικού προγράμματο Μεταρρυθμίσεων. Δεύτερη προτεραιότητα, να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στην πίστη, στι πιστώσει. Να ελευθερώσουμε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για να υποστηρίξουμε του εργοδότε και να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Οι πρόσφατε πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βοήθησαν πολύ για να αποφύγουμε πιστοτική κρίση και εμβάθυνση περαιτέρω τη ύφεση. Τρίτη προτεραιότητα είναι η ενιαία αγορά. Είμαστε αποφασισμένοι να την εκμεταλλευτούμε περισσότερο, οριστικόποιώντα την ψηφιακή αγορά και την ενεργειακή αγορά. Οι προτεραιότητες θα πρέπει να προωθούν μέτρα που κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ε, αποφασίσαμε να ανοίξουμε τις αγορές, η επιστροφή της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στις ε, Επιχειρήσει. Όπω συνέβη το 2009 μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και η μείωση που έγινε πρόσφατα των επιτοκίων μπορεί να ενισχύσει τι εξαγωγέ. Όλα αυτά βοηθούν. Αλλά βραχυπρόθεσμα όμω. Ο σκοπό είναι να υπάρξουν προοπτικέ και να υπάρξει ελπίδα μέσω των αποφάσεων του Συμβουλίου που έγινε πρόσφατα και αυτού που θα γίνει το Μάρτιο και τον Ιούνιο. Τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι και εμεί, αλλά και η Δανέζικη Προεδρία να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα για τη συνθήκη. Ε, σας ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερως, το ξέρω. Και κλείνει ένα κεφάλαιο το οποίο δημιούργησε πολλές συζητήσεις για δύο περίπου χρόνια. Όπως είπα, πολλές φορές εδώ στην ε, Ολομέλεια, από την εκκίνηση του ευρώ είχαμε πολλά προβλήματα και αυτή η συνθήκη είναι ένα στοιχείο των μεταρρυθμίσεων για την οικονομική διακυβέρνηση που έχουμε πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταρρυθμίσεις που αφορούν και τις ευθύνες αλλά και την αλληλεγγύη και προωθούν την αλληλεγγύη και που αφορούν το πακέτο των έξι μέτρων που είναι η ραχοκοκαλιά της νέας δομής διακυβέρνησης που προωθούμε. Αυτή η συνθήκη θέλει περισσότερη ανάληψη ευθυνών και καλύτερη υποπτία. Κάθε χώρα που την προσυπογράφει δεσμεύεται να ε, ε, βάλει στην νομοθεσία της κάποια μέτρα που ε, δημιουργούν τροχοπέδι στο χρέος και ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης θα εξασφαλίσει αυτή τη συμμόρφωση. Το να υπάρξει αυτό ε, θα ενισχύσει την αξιοπιστία της συνθήκης. Είναι σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αποτελεί ένα βασικό βήμα για να δημιουργήσει μια, να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομική και χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και θα υπάρξει δημοσιονομική βιωσιμότητα, θα, θα μειωθεί το κρατικό χρέος και θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει αυτοέλεγχος και αυτό δείχνει την μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να αποφύγουμε τα υπερβολικά ελλείμματα και τα υπερβολικά χρέη. Επίσης, η συνθήκη αλλάζει την πλειοψηφία που απαιτείται για να ξεκινήσει η διαδικασία υπερβολικού χρέους. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει με, με, την... τα μέτρα, τα έξι μέτρα, το six pack το λεγόμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι μια δέσμευση για λιτότητα. Αλλά είναι μία δέσμευση για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες ε, δαπάνες, αλλά όχι να αυξήσουμε το χρέος. Αυτό σημαίνει ε, όλο και περισσότερες δημόσιες δαπάνες ε, έτσι για την, ε, ξοδεύονται μάλλον για την εξυπηρέτηση του χρέους παρά για τις δημόσιες επενδύσεις. Το υπερβολικό ε, κρατικό χρέος είναι απειλή για το κοινωνικό μας μοντέλο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ήθελα να αλλάξουμε αυτά, όπως και εσείς θα θέλατε, να μην υπάρχει μια χωριστή συνθήκη, αλλά να κάνουμε αλλαγή στις σημερινές ε, συνθήκες. Αλλά δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία, η ομοφωνία μάλλον. Επομένως έπρεπε να προτάξουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος αυτές οι διατάξει να είναι όσο τον πιο κοντά στις σημερινές συνθήκες. Δεν δημιουργούμε ε, ένα χωριστό, μια χωριστή οργάνωση, αλλά δημιουργούμε τα μέσα για να ενισχύσουμε την ένωσή μα. Το ίδιο και με το, και με το σύμφωνο Europlus. Και ελπίζω ότι έτσι θα εσωματωθεί η συνθήκη αυτή, η νέα συνθήκη στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι εγώ προσωπικά δεσμεύτηκα να κρατήσουμε την Ένωση ως τον πιο α, συμπαγή, αναγνωρίζοντας ιδιαιτερότητες της Ευρωζώνης. Οι χώρες μας, επικυρώνοντας αυτή τη συνθήκη, θα συμμετάσχουν σε συνόδους κορυφής της ζώνης του Ευρώ, όπου συζητούνται οι βασικές αποφάσεις για το ευρώ και όπου η εφαρμογή της συνθήκη και συζητούνται και οι δεσμεύσεις των συμβαλωμένων μερών. Και βλέπω ότι σχεδόν όλες οι χώρες θα υπογράψουν τη συνθήκη. Θα τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν και μόλις ε, την επικυρώσουν 12 χώρες του ευρώ. Ο Χέλμαντ Μπροκ, ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, και ο κύριος Χόφστατ βοήθησαν ως εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου ε, σε αυτή την προσπάθεια. Τους ευχαριστώ. Η επιμονή του Κοινοβουλίου μαζί με άλλους για μια συνεπή στάση σε σχέση με τις απέναντι στις σημερινές συνθήκες βοήθησε ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής συνθήκης. Πέρα από αυτή τη συνθήκη για, για το δημοσιονομικό σύμφωνο, επίσης Έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα που θα υπογραφεί αυτή τη βδομάδα, ούτω ώστε να τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2012. Η έγκαιρη θέση σε ισχύ αυτού του βασικού μηχανισμού ανάσχεση του χρέου θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να μην περάσει η κρίση από τη μια χώρα στην άλλη. Ε, στις, το Μάρτιο, του 22, 22 ε, Μαρτίου του 2011 σας τα είχα πει όλα αυτά. Εν συνεχεία θα επαναξιολογήσουμε την επάρκεια των πόρων υπό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε πέντε εβδομάδες από τώρα. Και τέλος, κάτι που δεν ήταν επίσημα στην ημερήσια διάταξη, το συζητήσαμε. Θέματα εξωτερικής πολιτικής για το πώς Λαμβάνοντα υπόψη ε, τα συμπεράσματα της 23ης Ιανουαρίου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίσης, επικυρώσαμε τα πορίσματα των Υπουργών Εξωτερικών για το εμπάργκο στο Ιράν, στο Ιράν και επίσης καταδικάζουμε τη, τη βία του, του καθεστώτος της Συρίας και θέλουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η βία. Αυτά είναι καλά παραδείγματα μετά την κοινή δράση μα ε, για τη Λιβύη στα πλαίσια της ε, κοινή εξωτερικής πολιτική. Αυτά έχω να σας πω κυρίε και κύριοι. Βήμα-βήμα προχωρούμε για την οικοδόμηση μια οικονομική και νομισματικής ένωσης. Πιο αργά από ό,τι περιμέναμε, αλλά κάθε φορά υπάρχει μια ευρεία συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό συνέβη και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας. Έγιναν κάποια σημαντικά βήματα για το δρόμο πώς προς περισσότερη Ευρώπη. Ευχαριστούμε. ο Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Θα ήθελα να εμπιστήσω την προσοχή σας σε δύο πτυχές του ατύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Δευτέρας. Πρώτα απ' όλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πρώτη φορά ε, έκανε ένα σημαντικό βήμα στο να αναγνωρίσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πως δεν αρκεί μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η πειθαρχία με το να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και άρα η Κομισιόν ασχολήθηκε με τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες μας, την απασχόληση και την ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει συχνά με το Κοινοβουλίο μα και ξέρω πω υποστηρίζετε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βασίζεται στη στρατηγική τη Ευρώπη 2020. Βεβαίω χρειάζονται και άλλα βήματα και θα συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με την αποφασιστικότητα της ε, Κομισιόν να διατηρηθεί ο ρόλος της κοινοτικής μεθόδου και των θεσμικών οργάνων της κοινότητας στη νέα συνθήκη. Περνάμε σε μια νέα φάση οικονομικής διακυβέρνησης βασισμένη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όπου αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη πως ακόμα και ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας όπως η απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο λόγω του μεγάλου βαθμού αλληλεπίδρασης των οικονομιών μας. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα μόνο σε εθνικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας υπάρχει σαφώς μια ευρωπαϊκή διάσταση. Η εθνική και η περιφερειακή μάλιστα δράση πρέπει να στηριχθεί και να συμπληρωθεί από ευρωπαϊκή δράση. Τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης προφανώς δεν έχουν τελειώσει, μας περιμένει μακρύς δρόμος για την ανάκαμψη. Τονίζω την ανάγκη να συνεχίσουμε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, αυτή την οποία δηλαδή παρουσίασε η Κομισιόν στον οδικό της χάρτη πέρυσι τον Οκτώβρη. Από αυτή τη σκοπιά, σημαντικό ήταν οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων να συμφωνήσουν με την πρότασή μας να διασφαλίσουμε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να τεθεί ενισχύ ήδη τον Ιούλιο του 2012. Όπως συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο, το Μάρτιο θα αξιολογήσουμε ξανά την επάρκεια των πόρων του EFSF και του ESM. Ένα βασικό μήνυμα που προέκυψε από τη συζήτηση αυτή της Δευτέρας ήταν η ανάγκη να κάνουμε πολύ περισσότερα για να απελευθερώσουμε την δύναμη της ενιαίας αγοράς, το στολίδι του στέματος της Ευρώπης. Συμφώνησαν λοιπόν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν και την ιστορική ψηφιακή αγορά μέχρι το 2005 και ελπίζω να εγκρίνεται αυτό το πακέτο τους ερχόμενους μήνες με τη βοήθεια της Προεδρίας της Δανίας. Και ξέρουμε όλοι πόσο αποφασισμένη είναι η Δανική Προεδρία για όλα αυτά. Η ενιαία αγορά μπορεί να βελτιώσει το, βέλτιο, το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις μας, αλλά θα δημιουργήσει και τις καλύτερες θέσεις Εργασία ε, μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δημιούργησαν το 80% των νέων θέσεων εργασία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία μα. Και πρέπει να τι βοηθήσουμε να συνάψουν εμπορικέ συμφωνίε εκτό Ευρώπη. Το Δεκέμβρη που μα πέρασε προτείναμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία ω εγγυήσει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίση προτείναμε πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα οποία θα ήθελα να σα παρακαλέσω να υιοθετήσετε. Ζήτησα λοιπόν Δευτέρα να είναι ακόμη πιο φιλόδοξη η αρχηγή των κρατών και κυβερνήσεων στην περιστολή τη γραφειοκρατίας. Έκανα λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη τάση. Κάθε κράτο μέλο θα προετοιμάσει ένα εθνικό σχέδιο απασχόλησης ειδικά για τους νέους για να φροντίσει πως όλοι οι νέοι θα έχουν ή δουλειά ή η κατάρτιση εντός τεσσάρων μηνών από όταν τελειώνουν το σχολείο ή τη σχολή τους. Απίθυνα λοιπόν επιστολές ε, ειδικά στις χώρες οι οποίες πλήττονται ε, από την ανεργία των νέων. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε 22 δισεκατομμύρια από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να βελτιώσουμε τι πιθανότητε απασχόληση στην Ευρώπη. Να μεγιστοποιήσουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε, δηλαδή το Εράσμου, το Λεωνάρντο και το ΕΟΡΕΣ για την έβρεση θέσεων εργασία. Τα εθνικά σχέδια απασχόληση θα ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έτσι ώστε μέχρι το ΕΑΡΙΝΟ Συμβούλιο σε 6 εβδομάδε από τώρα να έχουμε συγκεκριμένε οδηγίε για όλα τα κράτη-μέλη. Επίση θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, σεβόμενοι τον ρόλο τους, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν ομαλώς τις στάσεις αυτές. Εγώ συναντήθηκα προσωπικά με εκπροσώπους τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ξέρω βεβαίως πως όλοι μαζί σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της ανεργίας. Ένα άλλο θετικό βήμα σε αυτό το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν το ότι ενέκριναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων την συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος της συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης της ΟΝΕ. Κάνουμε πρόοδο, όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν κάποιοι, αλλά κάνουμε πρόοδο προς μια δημοσιονομική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 κράτη-μέλη επίσης συμφώνησαν επί της ε, συνθήκης ε, συντονισμού και οικονομικής διακυβέρνησης, κατά το οποίο αποτελεί σημαντικό μέσο ανάκτησης της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης. Όπως ξέρετε, η συνθήκη αυτή δεν ήταν επιλογή της Κομισιόν, αλλά αποτέλεσμα της έλλειψης ομοφωνίας. Αλλά το γεγονός ότι 25 από τις 27 χώρες συμφώνησαν να υπογράψουν αυτή τη συνθήκη, νομίζω καταδεικνύει την αλληλεγγύη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ότι δεν υπάρχει διχασμός μεταξύ χωρών ευρώ και μη ευρώ. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων η Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο υπεράσπισε κάποιες βασικές αρχές, δηλαδή το ότι θα πρέπει να υπερέχει το ευρωπαϊκό δίκαιο, να διατηρηθεί ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, να συμπεριληφθούν όλα τα κράτη-μέλη και να ενσωματωθεί αυτή η συμφωνία στη συνθήκη της Λισαβόνας εντός πέντε ετών. Δεν υπάρχουν νέα θεσμικά όργανα λοιπόν, τα οποία θα μπορούσαν να εξασθενήσουν τον ρόλο της Κομισιόν. Τα συμβαλόμενα μέρη συμφώνησαν πως έχει κεντρικό ρόλο η Κομισιόν για την επίτευξη αυτών των στόχων και η κοινοτική μέθοδος και συμφώνησαν η συνθήκη να παραμείνει ανοιχτή προς όλους και να γίνει σεβαστή η κοινοτική μέθοδος. Τηρώντας την κοινοτική μέθοδο, η Κομισιόν έδρασε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω τη σημαντική συνεισφορά των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε πως ε, δράσαμε με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας όσον αφορά και την τροποποίηση του άρθρου 136 της συνθήκης. Σήμερα θα ήθελα να βεβαιώσω εξ ονόματος της ε, Κομισιόν το περιεχόμενο της επιστολής Όλη Ρεν προς Έλμαρ Μπρόκ και Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω πως ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο συμμετείχε ο Μάρτιν Σούλτς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην αρχή λοιπόν του Συμβουλίου έκανε μια σημαντική πολιτική παρέμβαση και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το ότι τήρησε τις αρχές οι οποίες είναι κοινέ στα δύο θεσμικά μας όργανα. Οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν πέρσι 23 Νοεμβρίου, το λεγόμενο διπλό πακέτο, πρέπει να μπουν στο πλαίσιο των συνθήκων, δηλαδή στα άρθρα 31 έως 36, καθώς επίσης και το ότι δεσμεύονται τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω δευτερεύουσα ε, νομοθεσία την οποία θα προτείνει η Κομισιόν. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής εγγύηση πως ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική διακυβέρνηση θα διασφαλιστεί μέχρι αυτή η νέα συνθήκη να ενταχθεί στις συνθήκες της Ένωσης. Μάλιστα, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά στις τρέχουσε προκλήσεις χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. συνεργασία μεταξύ των εθνικών δημοκρατιών και τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, η οποία βεβαίω αντιπροσωπεύεται από το κοινοβούλιο σας, μας δίνουν την απαραίτητη νομιμότητα να πάρουμε τις αποφάσεις οι οποίες είναι απαραίτητε για την ευημερία τη Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή για την ομάδα του ΕΛΚ. Ο συνάδελφο Ντόλ, τέσσερα λεπτά έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, αναλέθησαν οι ευθύνε ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράφοντας συνθήκη και επιθέμενοι στην, στα προβλήματα που υπήρχαν. Κατέδειξαν τη δυνατότητά τους να βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις στα ευρωπαϊκά προβλήματα. Ακόμα και αν δύο κράτη-μέλη προτίμησαν να μείνουν σόλο, θα λυπηθούν γι' αυτό στο μέλλον. Αυτή τη έχω τρει επιθυμίε. Η πρώτη είναι η συνθήκη να επικυρωθεί το γρηγορότερο δυνατό. Η δεύτερη να εφαρμοστεί το γρηγορότερο δυνατόν. Και η τρίτη αυτή η συμφωνία να ενσωματωθεί πλήρω στο ε, δίκαιο τη Ένωση, όπω το ζήτησε και το Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι, η οικονομική κρίση μα υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε τι συνήθειέ μα. Μα υποχρεώνει να σεβαστούμε του κανόνε, του προφανώ αλλά το δύσκολο να εφαρμοστούν για τη δημοσιονομική ισορροπία. Έχουμε την υποχρέωση να μειώσουμε τα εθνικά ελλείμματα που οφείλονται συχνά σε περιφερειακά και τοπικά ελλείμματα αλλά εφόσον η αποφάση για τη συνθήκη είναι ακριβής, εκείνες όμως για την ανάπτυξη δεν μου αρκούν. Γιατί το να καταπροωθούν τα ελλείμματα και να προωθηθεί η ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου νομιμίσματος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ενέργους κυρίως. Δύο τρόποι υπάρχουν να ξαναβρεθούμε την ανάπτυξη. Η μία τεχνητή και χωρίς αύριο, η άλλη δομική, άρα μόνιμη. Η πρώτη είναι να γίνει η ανάπτυξη μέσα της δαπάνης. Αυτό έγινε χρόνια και χρόνια και βλέπουμε που μας οδήγησε. Χωρίς να σκεφτούμε ότι σήμερα οι δαπάνες de facto είναι περιορισμένες, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να επιστρέψουμε τα, τα δανεικά και όχι να ξαναδανειμόμαστε. Η δεύτερη είναι εκείνη που έχει κατά νου το ΕΛΚ, δηλαδή η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική. Αυτό μπορεί να γίνει, αγαπητέ Μανουέλ Μπαρόζο, ε, προωθώντας τέλο την εσωτερική αγορά. Όλα τα κείμενα έχουν εγκριθεί εδώ και πολύ καιρό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να μας κοινοποιήσει το γλυγορό των ετών ποιο δεν εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες και να τους υποχρεώσει να την εφαρμόζουν πώς είναι η υποχρέωση της Κομισιόν που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Και η Γαλλία ίσω και η Γαλλία δεν από καμία εξαίρεση αγαπητοί φίλε Ε, κάθε Ευρωπαίος πρέπει να ξέρει ποιος, ποια χώρα παρεμποδίζει την εσωτερική αγορά. Αυξανώντα την ανταγωνισμό μα, μπορούμε να μειώσουμε και την επιβάρυνση των ε, επιχειρησιών και μειώνοντα ε, εκείνη ε, την επιβάρυνση που πλήττει την ανταγωνιστικότητα επί επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εκείνα τους πόρους από τα κοινωτικά ταμεία που δεν χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε σε κοινά σχέδια που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και σε απασχόληση. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με ε, επενδύσεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη και με ε, εξέταση εκείνων των ε, δημοσίων δαπανών που δεν οδηγούν σε ανάπτυξη. Μια που το 1 τέταρτο της νεολαίας είναι σε ανεργία, οφείλουμε να τους βοηθήσουμε και να μπορέσουν να προσανατολιστούν στο σύνολο της Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Τόλ. Ο Σάρφος Σόβοντα για την ομάδα του 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε και ακούμε πως η ενεργεία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 13 χρόνια. Και τι μας προσφέρει εδώ πέρα το Συμβούλιο, μια συνθήκη εκτός κοινοτικής ε, μεθόδου και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς και πότε θα τεθούν ενισχύ και η κακοφωνία βεβαίως συνεχίζεται. Σκεφτείτε πως υπήρχε επίσης μία παράξενη ιδέα να οριστεί ένας επίτροπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση από κάποιο κράτος μέλος για την Ελλάδα. Το κόμμα μου είναι οπωσδήποτε κατά το να υπονομεύσουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα μέσω του ορισμού ενός τέτοιου επιτρόπου. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Η κατάσταση επίσης είναι αποτέλεσμα του πώς έχει παρεξηγήσει η κυρία Μέρκελ τον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας. Βεβαίως η Γερμανία είναι μια μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη, αλλά θα πρέπει να έχει τη δύναμη να συμβιβάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να τη διχάζει. Και όταν η Handelsblatt, η οποία δεν είναι και καμιά δεξιά ε, ε, αριστερή εφημερίδα, γράφει πως δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος για την Ευρώπη, κάτε πάει καλά εδώ πέρα. Εάν μου επιτρέπετε λοιπόν να πω Κάτσε, η κυρία Μέρκελ θα πρέπει να δει τους ε, εταίρους της. Αν δούμε και τον ε, το μελλοντικό πρόεδρο της Γαλλίας, τον Φρανσουά Ολάντ. Ναι, ναι, τον... τον υποστηρίζουμε όπως υποστηρίζουμε και την ε, πρόθεσή του να επαναδιαπραγματευτεί αυτή την συνθήκη. Και ούτως ή άλλως δεν θα βοηθήσει η κυρία Μέρκελ τον προεκλογικό αγώνα του ε, κυρίου Σαρκοζή. Αλλά εάν δείτε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Πορτογαλία, δεν βοηθάνε αυτά τα συμπεράσματα ούτε τις χώρες, ούτε κανέναν άλλον να οδηγηθεί σε περισσότερη σταθερότητα. Πρέπει να φύγουμε και να απομακρυνθούν αυτές οι χρηματαγορές, να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα μέσα ενός φόρου στις ε, συναλλαγές τους και να εξοδευτούν τα λεφτά εκεί ακριβώς όπου τα χρειαζόμαστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πράγματι υπήρξαν κάποια θετικά στοιχεία. Επιτέλους ασχολήθηκε το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό με την ανεργία των νέων, αλλά μπορείτε να μου ε, εξηγήσετε γιατί για το έλλειμμα υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι και κυρώσεις και δεν υπάρχει τίποτα για την ανεργία των νέων. Όχι, είναι μια ανισορροπία η οποία είναι απαράδεκτη. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μπούζεκ για το ότι πίεσε να συνδιαπραγματευτεί και το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει κάποια μεγάλα λάθη. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο, τον κύριο Μάλτιν Σούτς. Πραγματικά είπατε τις κατάλληλες λέξεις με το σωστό τόνο για να ακουστείτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Κομισιόν. Έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το λάθος που γίνεται με αυτή τη συνθήκη να γίνει κανόνας. Θα πρέπει να παραμείνει εξαίρεση. Και εδώ πέρα... Ε, θα πρέπει νομίζω να ενισχύσουμε και να μην το μετανιώσουμε τον ε, Μάρτιν Σούλτς με την ε, ψήφο μας για να έχει μια ισχυρή φωνή από εδώ και μπρος στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σφόποντα. Ε, λόγω του περιεχομένου των ε, τελευταίων ε, λέξεων, σε άφησα μιλήσει λίγο παραπάνω. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Λάμπζορφ. Παρακαλώ. Ναι, αγαπητέ Σβόμποντα. Συμφωνείτε πως οι ίδιες χώρες οι οποίες αυτοί αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες με το χρέος είναι επίσης οι ίδιες χώρες με την υψηλότερη ενεργεία των νέων και πως ε, ακριβώς ε, το ζήτημα της ε, απασχόλησης είναι θέμα των χωρών αυτών και των επιχειρήσεων βεβαίως που θα πρέπει να φροντίσουν να απασχολήσουν τους νέους. Δεύτερον, παρακαλώ αφήστε τους Γάλλους πολίτες να εκλέξουν μόνοι τους πρόεδρο. Ευχαριστώ. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ναι. Στη μία ερώτηση που να θα ψηφίσουν οι Γάλλοι ό,τι θέλουν και από εκεί πέρα ε, κάποιος που ξέρει τι θα κάνει και έχει βρει μια ιδιωτική δουλειά για μετά έχει αναγνωρίσει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκτός αυτού θέλω να σα πω ότι για μένα και την ομάδα μου η ανεργία είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Και η ανεργία των ένων είναι τόσο ψηλή γιατί κανένας δεν σκέφτηκε ότι καμιά φορά θα πρέπει να υπάρχουν ενεργά μέτρα. Κοιτάξτε τις χώρες που έχουν χαμηλή ανεργία. Ελάτε στην Αυστρία, ελάτε. Έχουμε την πιο χαμηλή ανεργία, γιατί κάνουμε πολλά. Και το λέω και στους συναδέλφους για προάλληλη. Είναι ντροπή η ανεργία. Ε, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, διακόπτη τον ομιλητή. Das Wort hat nun für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten Herr Verhofstadt. Για την ομάδα του Yes, uh, chairman. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε μια σύνοδος κορυφής τη Δευτέρα για την ανάπτυξη και για την ανάπτυξη και απασχόληση. Κατά τη γνώμη μου, όπως είπε και ο κύριος Ντόλ, παρήγε λέξεις κυρίως. Εφτά σελίδες ε, λέξεις και εφτά σελίδες καλές προθέσεις. Τώρα είμαστε το μέσο της κρίσης. Δεν χρειαζόμαστε 7 σελίδες λέξεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πράξεις. Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Να σας δώσω τρία παραδείγματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Μόνο. Το πρώτο. Το Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένα μεγάλο εργαλείο για την ανάπτυξη στην Ευρώπη για πάνω από ένα χρόνο έχει μπλοκαριστεί η εισαγωγή του. Γιατί? Γιατί οι μεγάλες χώρες προς το παρόν δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την έδρα του οργανισμού που ασχολείται με αυτά τα διπλώματα ευρεσίγνεχνίας. Για την έδρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάτι που είναι γελίο. Για να μην πω και δραματικό παράλληλα. Γιατί στο μεταξύ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας πληρώνουν 8 φορές περισσότερο για την προστασία των καινοτομιών τους από ό,τι πληρώνουν οι Αμερικανοί ομολογοί τους. Απευθύνομαι στον πρόεδρο του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία τελικά. Γιατί οι Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει οι ηγέτες, αφού δεν συμφωνούν αυτές τις τρεις χώρες, ας βάλουμε την έδρα στις Βρυξέλλες. Όπως το κάναμε, κύριε Κονπεντίτ, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων το 2001 είναι ντροπή να έχουμε μια σύνοδο κορυφή του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε να δρομολογήσουμε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Είναι τα ομόλογα έργων. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει αυτό το περίφημο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Για χρόνια το συζητάμε. Το ερώτημά μου είναι, γιατί να μην αρχίσουμε αύριο με αυτά τα έργα με αυτά τα ομόλογα έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει δηλαδή να περιμένουμε δύο χρόνια να κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις στο Συμβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα. Και να σας δώσω κι άλλο παράδειγμα, ένα τρίτο παράδειγμα. Τα τεράστια ποσά αχρησιμοποιητών κονδυλίων από τα διαρθωτικά ταμεία και άλλα ταμεία. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κανονισμό πάρα αυτά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν βάλετε ένα ευρώ από τα διαρθωτικά ταμεία, χρειαζόσαστε επίση ένα ευρώ από τη χώρα. Και οι χώρε δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να συγχρηματοδοτήσουν. Μιλάω για την Ελλάδα, α πούμε. Μιλάω για την Πορτογαλία. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε πάρα αυτά, τώρα, εδώ και τώρα, να αλλάξουμε τον κανονισμό. Και πάρα αυτά να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρησιμοποιητά μη δαπανηθέντα κονδύλια για τι χώρε που βρίσκονται σε ύφεση, όπω η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Πράξει και όχι λόγια. Όχι 7 σελίδε από λέξει, λέξει, λέξει. Τέλος, άλλο πρόβλημα σήμερα. Υπαρξιακής φύσης έχουμε εδώ πέρα σε αυτή την ευρωκρίση. Έχουμε τη νέα συνθήκη, ωραία, την εξασφαλίσαμε. Ωραία, τώρα έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία, έχουμε τα... το πακέτο των 6 μέτρων, των 2 μέτρων, τη νέα συνθήκη. Πώ θα ασχοληθούμε με τα ακόμα υψηλά επιτόκια, ακόμα και μετά την παρέμβαση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε χώρε όπω Ισπανία και η Ιταλία. Όλοι σας ξέρετε ότι τα επιτόκια των 6% είναι μη βιώσιμα για την Ιταλία. Ο κύριος Μόντι, ό,τι και να κάνει με τις αποφάσεις του, δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα επιτόκια και η Ιταλία δεν πρόκειται να κάμψει με αυτά τα επιτόκια των 6%. Ήδη, συνάδελφοι, έχουμε βάλει πάνω από ένα 3 ευρώ για να καταπολεμήσουμε αυτή την, την κρίση. Από τα λεφτά των φορολογουμένων. Και όμως δεν έχουμε βγει από το τούνελ. Και ο λόγος είναι γιατί παίρνουμε, ότι παίρνουμε με ημίμετρα. Χρειαζόμαστε διαφορετικές λύσεις για αυτή την κρίση. Και κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνει το χρέος να το αντιμετωπίσουμε από κοινού με πειθαρχημένο τρόπο. Οι πέντε σοφοί οικονομολόγοι αυτό πρότειναν για να υπάρξει διαφυγή από την κρίση. Συμπέρασμα, Πρόεδρε ένα μήνυμα προς τους Γερμανούς ε, φορολογούμενους. Αυτοί που έχουν τα ομόλογα ε, λαμβάνουν λιγότερα επιτόκια. Εγώ λέω, ας δημιουργήσουμε ένα ταμείο για να προχωρήσουμε όλα αυτά τα μέτρα και να ξεφύγουμε από τα απλά ευχολόγια. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χάμς ε, για την ομάδα των Πρασίνων. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Μετά τη κορφή διάφασα στι εφημερίδε ότι ορισμένοι θεώρησαν καταπληκτικό επιτεύγμα αυτή η διάσκεψη κορυφή και το σύμφωνο σταθερότητα. Αν δούμε όμω ακριβώ τι έγινε, θα λίγα εγώ σε άλλο αποτέλεσμα. Γιατί έλεγε Έχουμε μια συνθήκη. Προετοιμάζεται ακόμα, θα δούμε που θα καταλήξει. Μια συνθήκη η οποία έχει σαν στόχο οι ισχύουσες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρηθούν. Και αυτή η συνθήκη τοποθετείται εκτός των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και καταφέρνουν και η δημοκρατία να μείνει εκτός των συνθήκων με την αυτή συνθήκη. Εάν αυτό είναι το καταπληκτικό επίτευγμα, τι να σας πω. Κύριε Ρόμπο ή κύριε Μπαρόζο, αν μπορώ να σας λάβω σοβαρά η υπόψη. Εγώ σας θεωρώ για πολύ πιο σοφούς πολιτικά από εκείνα που μας είπατε σήμερα για τελευταία αυτή άτυπη σύνοδο κορυφής και τα αποτέλεσματά της. Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ε, πολιτική κομμωδία. Δεν νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν οι πολίτες τόσο πολύ γι' αυτό. Όσο πάει οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι τους εξαπατά το, η διάσκεψη με την κομμωδία αυτή που παίζει. Το μεγάλο πρόβλημα κατά γνώμη είναι ότι η ανάλυση λέει ακριβώς ότι το δημόσιο χρέος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κρίση. Και όσο και αν προσπαθώ εγώ να κατανοήσω την ανάλυση της κρίσης, δεν καταφέρνω στο ίδιο αποτέλεσμα να φτάσω. Αλλά το ότι τσακωνόμαστε εδώ και χρόνια για τους προπολογισμού μας και πώς θα σου το εξηγιάσουμε, αυτό επιδεινώνει αυτή την ιδέα της κρίσης. Αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης της ύφεσης για τις χώρες αυτές ε, που βρίσκονται σε κρίση. Μας λέτε διάφορα εδώ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτά όλα έχω δει ότι δεν λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Ξέρω να διαβάζω, ξέρω να μετράω και να κάνω υπολογισμούς. Πού είναι αυτές οι θέσεις απασχόλησης επιτέλους. Πού είναι τα χρήματα στα οποία θα βασιστούν οι δηλώσεις σας αυτές. Εγώ δεν το βρίσκω να υπάρχει τίποτα. Ας ρίξει κανένας μια ματιά στην Ελλάδα, μια ματιά στην Πορτογαλία. Ο κίνδυνος μετα... αναμετάδοσης θα πρέπει να ξέρει ο καθένας τι χρειάζεται η Ελλάδα. Έναν επίτροπο για εξοικονομήσεις, άλλον Ευρωπαίο τεχνοκράτη δηλαδή που έχει εντάξει εκεί μια τεχνική, τεχνητή κυβέρνηση στη χώρα αυτή. Θέλουν άλλον επίτροπο από πάνω. Χρειάζονται επιτέλους μια ειλικρινή ανάλυση οι Έλληνες και μια αναγνώριση του προγράμματος κατά τη ύφεσης για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Χρειάζεται στην ενέργεια, στην υποδομή νέα προγράμματα. Είναι έτοιμα τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν επίτροπο για οικονομίες, για λιτότητα, αντί να συζητάμε με τους Έλληνες για την Ελλάδα τη αύριο, αντί να εθαρρύνουμε τους Έλληνες. Αυτό πραγματικά είναι το να δει τη όλη τη συζήτηση, ότι έτσι μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και η Ελλάδα. Ντράπηκα πραγματικά για αυτά που άκουσα και διάβαζα κύριε Φαν Και τελειώνοντας τι γίνεται με τις χώρες που είναι ακόμα εκτός ευρώ. Πρέπει κάποια στιγμή να το εξετήσετε μεταξύ μας να το δούμε αυτό. Πώς θα το, ε, θα το εξηγήσετε. Οπωσδήποτε δεν είμαι η καλύτερη φίλη του Ντονάλτους. Όχι. Αλλά όταν πρόκειται για την Ευρώπη και όταν θέλουμε να σκεφτούμε το σύνολο και όχι τα μικροσυφέροντα τούτου και του άλλου των πλουσίων χωρών της Ένωσης, όταν εξετάζουμε το σύνολο Μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από τον Ντονάλτο στο να τσακωνόμαστε μαζί του για το ρόλο του. Εδώ πραγματικά είχαμε τον Ναδίλ της Ευρωπαϊκής Ένωση. Καταπληκτικό αποτέλεσμα είναι κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. ευχαριστώ κυρία Χάμς. Για το ομάδα της ΕΡ, ο συνάδελφος Κέλενεν. Τρία λεπτά. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία σήμερα στο Κοινοβούλιο πως ακόμα και αν υιοθετηθεί και εγκριθεί αυτό το σύμφωνο, κάτι το οποίο δεν ε, είναι βέβαιο, αν έχει δίκιο ο κύριος Φόβοντα, δεν θα λυθεί η κρίση. Και ως ε, συντηρητικός, ως μπροστά δημοσιονομικά, εγώ θα έπρεπε να χαίρομαι για το ότι πλέον θα γραφτεί σε εθνικούς νόμους και συντάγματα κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι πως η δυνατότητα των ψηφοφόρων να ψηφίσουν μια κεντσιανή πολιτική καταργείται. Κάνουμε παράνομο το σοσιαλισμό, κύριε Πρόεδρε. Και αυτό το σύμφωνο καθιστά άκυρες τις εκλογές σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Ως συντηρητικός λοιπόν της ελεύθερης αγοράς που θαυμάζω πολλά πράγματα στο γερμανικό μοντέλο δημοσιονομικής και μονεταριστικής πειθαρχίας δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο την ισχύ του νόμου αλλά και των επιχειρημάτων. Πρέπει να δείξουμε πως η λιτότητα δεν κρατάει για πάντα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Αλλά εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγει κάποια χώρα από το ευρώ, τότε μπλοκάρουμε αυτό το τούνελ. Καταδικάζουμε τις χώρες σε πολλά χρόνια φτώχειας και μετανάστευσης. Δεν θα έρθει ανάκαμψη στην Νότια Ευρώπη μέχρι να έχουν οι χώρες δικά τους νομίσματα. Και βεβαίως δεν μπορούμε να τους μιλάμε για λιτότητα εάν δεν την εφαρμόζουμε και οι ίδιοι. Φανταστείτε πώς φαίνεται η ευρωπαϊκή ε, το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο με τα γεύματα, τους διάφορους παρατρεχάμενους σε ένα δημόσιο υπάλληλο με όλες τις περικοπές που έχει υφωστεί. Σκεφτείτε πώς νιώθουν οι φορολογούμενοι όταν κάνουμε οικονομίες και πληρώνουμε περισσότερο στον προπολογισμό της Ένωσης. Η ομάδα μου βεβαίως είναι υπέρ της εσωτερικής αγοράς και θα συνεχίσουμε να είμαστε υπέρ της επέκτασης και των υπηρεσιών και να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Θα συνεχίσουμε να θέλουμε καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της εσωτερικής αγοράς και βέβαια το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς δεν έχει νόημα παρά μόνο να ανοίξουμε την αγορά μας στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί δηλαδή που υπάρχει ακόμα ανάπτυξη. Αλλά πολλά από αυτά είναι μέσω μακροπρόθεσμα. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εδώ και τώρα για να δείξουμε σε επιχειρήσεις πως είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Οπωσδήποτε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να καταργήσει τη διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων, να πάνε οι αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη και να καταργηθούν διάφορες οδηγίες ε, περί εγκυμοσύνης, χρόνου εργασίας και διάφορα άλλα εμπόδια εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις ε, απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό δεν γίνεται με ψηφίσματα. Εμείς οι ευρωκράτες και οι ευρωβουλευτές δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καμία θέση εργασίας. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εμποδίζουμε τους επιχειρηματίες να εφευρίσκουν, να φτιάχνουν και να πουλάνε πράγματα. Από εκεί προέρχεται η απασχόληση και η κοινωνική ασφάλιση. Όταν ήμουν νέος Ευρωβουλευτής υπήρχε κάτι το οποίο λέγαμε η ατζέντα τη Λισαβόνα που θα έκανε μέχρι το 2010 την Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου. Όπως τα λέει η Σάρα Πέιλιν, πώς ε, τα πήγαμε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπίσκι για την Γκουε για δύο λεπτά. Ε, Πρόεδρε, η απελευθέρωση των οικονομικών αγορών οδήγησε σε μια ανάπτυξη των αγορών αυτών που μέχρι στιγμής δεν ελέγχεται. Μόνο ζωσπαστικά μέτρα για την αποτροπή των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων στις αγορές αυτές μπορούν να αποτρέψουν και να περιορίσουν την κρίση. Από την άλλη μεριά με την έγκριση της δημοσιονομική Συμφωνίας βλέπουμε επιδείνωση της μονομερούς αυτής ε, οργάνωσης και προσανατολισμού αυτή η γραμμή της μείωσης των χρεών και των ε, δημοσίων δαπανών την απορρίπτει δική μου πολιτική ομάδα. Είναι κάτι που επικρίνεται και από το Εθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Βος λέει ότι αυτή η πολιτική θα οδηγήσει την Ευρώπη σε αποπληθωριστική πτώση προς τα κάτω. Η συμφωνία προβλέπει περιορισμό των χρεών και θα πρέπει να επιβληθεί αυτό με την έγκριση και υιοθέτηση του εθνικού δίκαιου. Αλλιώ θα υπάρχουν κυρώσει από την Κομισιόν και το δικαστήριο αυτό είναι παράλογο, αντιδημοκρατικό. Γιατί τα κράτη χάνουν τη δημοσιονομική τους ε, κυριαρχία. Από την άλλη μεριά επίσης είναι απαράδεκτο η αλληλέγγυη βοήθεια για χώρες που βρίσκονται προ... που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα να συσχετιστεί με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Γιατί έτσι υποσκάπτεται η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θυσιάζεται στο βωμό των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Θα πρέπει να έχουμε μια συμφωνία για υφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. Θα χρειαζόμαστε δημόσια προγράμματα για επενδύσεις για το περιβάλλον και την παιδεία. Κυρίως χρειαζόμαστε μια δημοκρατική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών. Θα πρέπει η συμβάση αυτή να εγκριθεί με ε, δημοψήφισμα. Ευχαριστώ κύριε Μπίς, κύριε Πρόεδρος. Για την ευθύ ο κύριος Φαράς έχει το λόγο. Well, Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ο Ντέβιτ Κάμερον μας έκανε να ανησυχήσουμε αλλά τελικά έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Τι έγινε με το βέτο, κανένας δεν το ασκεί. Ο κύριος Κάμερον μάλιστα τώρα υποστηρίζει αυτό το αφρικτό σύμφωνο που θέλει να καταστρέψει και να ταπεινώσει τα εθνικά κράτη τα οποία δεν πληρούν αυτά που λένε και δεν κάνουν αυτά που λένε οι Γερμανοί. Ένας υπουργός ε, Γερμανός είπε ότι θα πρέπει κανονικά να πάνε οι ευρωκράτες στην Αθήνα και να καταλάβουν εκεί ένα μεγάλο κτίριο για να βάλουν τάξη. Νόμιζα ότι ήταν αστείο, αλλά όχι, ήταν μια διαπραγματευτική θέση. Και τώρα τι πετύχαμε για την Ελλάδα. Είναι ε, μια διπλωματία με στραμμένο το όπλο προς τους Έλληνες. Κανένα δεν μπορεί να αρνηθεί σήμερα ότι η Ελλάδα είναι μια απικία. Αλλά όλα αυτά είναι τεράστια λάθη. Ε, η Ελλάδα δεν είναι μια επικουρική ε, εταιρεία που δεν τα πάει καλά και πρέπει να πάμε εμείς να την ε, ελέγξουμε. Είναι ένα έθνος με περηφάνεια, με ιστορία. Αυτοί εφήβραν και τη δημοκρατία μάλιστα. Και σήμερα έχουν τεράστια προβλήματα. Έχουν ανεργία των νέων ύψου 50%. Γιατί, κύριε Φανρόμπου, γιατί είναι στο ευρώ. Εσείς δημιουργείτε τη μιζέρια και την ε, ε, δυστυχία αυτής της χώρας. Και λέτε φλιαρίε περί δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αλλά τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Οι Έλληνε ταπεινώνονται και είναι σε φάση απελπισία. Και οι απελπισμένοι άνθρωποι κάνουν απελπισμένα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ελλάδα αν συνεχίσουμε αυτή την τρελή τροχιά. Κύριε Μπαρόσο, ξέρετε πολύ καλά ότι η δική σας χώρα είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, κύριε κύριος Μπρόντς. Για τους μη ταγμένους, για τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο κύριος Μπρόντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καμερών είπε ότι δεν θα περιποτήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από την εφαρμογή τη Εθνική Συμφωνία για την πολιτική. Φαίνεται τελικά όμως ότι υποσχέθηκε κάτι για κάτι που δεν μπορεί να αποτρέψει, αλλά πρέπει να το αποτρέψει. Το άρθρο 8 της ε, πρώτας συμφωνίας λέει ότι θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο 273 για να εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή και πραγματικά το άρθρο 273 λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να έχει δικαιοδοσία για οποιαδήποτε συμφωνία ε, μεταξύ κρατών αφορά την σύμβαση μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να βάλει πρόστιμα στα κράτη-μέλη αν δεν συμφωνούν. Επίσης, η δικαιοδοσία δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξετάσει υπερβολικά ελλείμματα των προπολογισμών. Το άρθρο 8 λέει ότι η Κομισιόν θα μπορεί να ξεκινήσει κάποιες δράσεις, αλλά αυτή, αυτό το σχέδιο συμφωνίας είναι μια συμφωνία που δεν μπορεί να το κάνει, γιατί το άρθρο 273 αναφέρεται σε διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών, όχι διαφωνίες με την Κομισιόν. Άρα η Κομισιόν φαίνεται ότι δεν έχει την ισχύ να ξεκινήσει εδώ μία δράση ενώπιον της δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι δεν έχει κανένα ρόλο η Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να λέει κατά πόσον συμβιβάζεται ή δεν συμβιβάζεται μια χώρα με τη συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί και πέρα. Ε, θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, χρειαζόστε μια νέα συνθήκη, η οποία θα πρέπει να συμφωνηθεί ομόφωνα. Θα ήταν ε, καταστροφικό για τη Βρετανία να συμφωνήσει με τέτοιο μηχανισμό, γιατί τελικά ίσως σήμερα είναι ει βάρο των χωρών τη Ευρωζώνη, αλλά μεθαύριο μπορεί να είναι και ει βάρο εμών. Συγγνώμη, δεν είδα την πλεκάρτα κάρτα σας. Ποιον θέλετε να ρωτήσετε. Ο κύριος Φάρατς μίλησε για Γκάουλάιτερ. Ως Γερμανός διαμαρτύρομαι να εξισώνεται τη δημοκρατική Γερμανία με την εθνικοσοσιαλιστική. Γι' αυτό θέλω συγνώμη από αυτόν τον άνθρωπο. Κανείς στο Βερολίνο δεν στέλνει Γκάουλάιτερ στην Ευρώπη. Αυτά είναι κηρύγματα μίσους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των, των Ευρωπαϊκών λαών. Πρέπει να το πάρετε πίσω και εσείς πρέπει να φροντίσετε να μην ξαναεπαναληφθεί αυτό το πράγμα. Κάποιοι θα έλεγαν. Και η μεγαλύτερη κυριακάτικη εφημερίδα χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αν θέλετε να μιλήσετε για μίσος, κοιτάξτε τι κάνει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Οι γερμανικές εφημερίδες βρίζουν τους Ιταλούς ότι είναι δειλούς, τους Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες και άχρηστοι. Οι δε ελληνικές και οι ιταλικές απεικονίζουν τους Γερμανούς ηγέτες με ναζιστικές στολές. Οπωσδήποτε. Το οικοδόμημα αυτό που νόημα είχε την ειρήνη και την αρμονία μας διχάζει και επαναφέρει τον εθνικισμό. Και αν υπήρχε μία χώρα στην οποία επιτέθηκα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παραδέχτηκα πως ο τρόπος στον οποίο, με τον οποίο συμπεριφερθήκαμε εμείς στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα δεν ήταν σωστός. Ο εθνικισμός ε, σε αυτή την αίθουσα ε, διαχέεται και από κάποιους οι οποίοι βάζουν ε, σημεούλες στα έδρανά τους νομίζω για να δείξουν από πού κατάγονται. Τέλος πάντων το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε. Das Wort hat der Kollege Το λόγο έχει ο συναλφός Μπρόκ. Καθίστε σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει ο κύριος Μπρόκ. Ich rufe Sie, jetzt, zur Ordnung. Setzen Sie sich hin. Σας καλώ σε τάξη. Παρακαλώ καθίστε. Κύριε Βουλευτά Φαράτσου, καθίστε παρακαλώ, αλλά θα σας πω να φύγετε από την αίθουσα. Ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Μπαρόζο και Φενρόμπο που ήρθαν εδώ και που βοήθησαν πραγματικά την ομάδα υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, θα σας πω, εμείς δεν θέλαμε αυτή τη συνθήκη, θέλαμε μια κοινωτική συνθήκη, αλλά λόγω της τάσης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν δυνατό αυτό, γιατί είχαν πει ότι δεν επιτρέπει να διακανονίσουμε την, οικονομικοπιστωτική αγορά. Εμείς θέλουμε να διακανονίσουμε για να μην μας καταστρέψουμε. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να απορρίψουμε αυτό που ζητούσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και άμα ακούω αυτούς τους κύκλους, να επανέρχεται η γλώσσα του παρελθόντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε ειρήνη, ευημαρία στην ε, ε, Ήπειρο αυτή που δεν είχαμε ποτέ. Δεν το επιτρέπω αυτούς τους κυρίους από ο κ. Φαράντ και άλλους να μου το καταστρέψουν. Αυτή η συνθήκη επιτρέπει να τραγουδήσουμε τα χρέη. Δεν ήταν δυνατό αυτό με τη σημερινή κοινοτική συνθήκη. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να παραμείνουν αυτά. Ότι όλα τα άλλα να υπάρχουν στην κοινοτική νομοθεσία. Και αυτό το πετύχαμε. Να ισχύουν δηλαδή οι κοινοτικοί κανόνες, να γίνονται όλα μέσα σε κοινοτικά πλαίσια και το δικαίωμα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κύριε Μπαρόζο, σας παρακαλώ γλίγορα να υπάρχουν τώρα προτάσεις πως θα γίνει κάτι τέτοιο συγκεκριμένο στην εφαρμογή της ε, Σύμβασης Ανάπτυξης γιατί η Ελλάδα και οι άλλες ε, χώρες δεν πρέπει να περιμένουν να δουν ότι κάτι γίνεται πραγματικά συγκεκριμένο χρειαζόμαστε, επιταρχία χρειαζόμαστε, ερωτικές αλλαγές στις χώρες αυτές θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες που υπάρχουν. Όταν βλέπω ότι υπάρχουν 16 δισεκατομμύρια στο λογαριασμό για την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν μπορεί να υποβάλει τα σχετικά σχέδια να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να τη βοηθήσουμε, περί αυτού πρόκειται κυρία Σφόποντα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε να ελέγχει τη δίκη της ώστε να μπορέσει να προωθήσει την αναπτύξωση. Η κυρία Μέρκελ είναι υπέρ της ε, πειθαρχίας, της ανάπτυξης και διορθωτικών αλλαγών. Εσείς ξεχάτε την πειθαρχία και καταστρέφετε το μέλλον των, υπερχομένων των ε, επερχομένων γενιών άμα ξεχνάτε την πειθαρχία. Η κοινοτική μέθοδος και ε, διασφαλίζεται και τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τη διπλή ε, αλληλεγγύη που θέλει και η κυρία Μέρκελ. Ο καθένας θα πρέπει να βοηθήσει αυτόν και πάνω σε αυτό θα τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η στρατηγική και παρακαλώ οι σοσιαλιστές να υπερψηφίσουν τον κύριο Σαρκοτζή να το υποστηρίξουμε αυτό. Ο Μητερό χρειάστηκε δύο χρόνια μέχρι να μπορέσει να ακολουθήσει τη γραμμή που ε, ακολουθήσε. Εάν εκλεγεί ο κύριος Ολό θα δείτε πώς θα γίνει δύο, μέρες, δύο εβδομάδες μετά που θα αναλάβει το έργο του. Θα αλλάξει ριζικά, αλλιώς θα καταστρέψει τη Γαλλία. Κύριε Μπρόκ, σα έδωσα συμπληρωματικά πάνω από ένα λεπτό, γιατί είσαστε ένα από ε, του επιτυχεί διαπραγματευτέ του σώματο. Αλλά. Ακούστε με, κύριε. Κύριε Μπρόκ, ακούστε με, σα παρακαλώ. Ακούστε με. Με όσα είπατε, οδηγήστε σε ένα κατακλυσμό μπλε καρτών. Ο κύριος Μάτλεν ήταν πρώτος. Μόνο σε εκείνο θα επιτρέψει να μιλήσει. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ξεκαθαρίσατε κάτι σημαντικό εδώ πέρα, γιατί μπορεί ο κύριος Μπρόκ να μας λέει πως ε, η Ευρώπη φροντίζει για την ε, ελευθερία, αλλά δεν είμαι πλέον τόσο σίγουρος. Θεωρείτε εσείς ε, κύριε Μπρόκ, πως είναι φυσιολογικό να τεθεί υπό εποπτεία μια χώρα χωρίς να ερωτηθούν οι κάτοικοί τη ή το να εκδώσουμε ευρωομόλογα χωρίς να ρωτήσουμε τους δικούς μας ψηφοφόρου εάν το επιθυμούν. Νομίζω πως έχουμε φτάσει στα όρια του δημοκρατικού εφικτού και τα έχουμε ξεπεράσει. Οπότε Ξεωρείτε λοιπόν πως θα πρέπει να μπορούν να εκφραστούν και οι Έλληνες και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί μέσω δημοψηφισμάτων για να μας πούν ποιο θέλουν αυτοί να είναι το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, πρώτα απ' όλα να διαπιστώσουμε πως κάθε χώρα πρέπει να τηρεί τους κανόνες τους πρέπει να γίνει αυτό. Όταν αποδέχεται κανεί του κανόνε και υπογράφει οι συνθήκε, πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόζονται. Δεν είναι τίποτα το διαφορετικό εδώ πέρα. Δεύτερον, όλα τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν θα περάσουν μόνο με αποφάσει των εθνικών κοινοβουλίων. Του γερμανικού, του εθνικού, του, του γερμανικού, του ελληνικού, του ολλανδικού. Πλην τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν συμμετέχει σε αυτή την αλληλεγγύη για την Ελλάδα. Αυτά προς τον κύριο Φαράζ για το πώς συμπεριφερόμαστε δέστε αυτούς λαούς. Το ότι θα μπορούσαμε δε να έχουμε κάποιον επίτροπο ο οποίος θα ασχολούνταν για όλες τις χώρες οι οποίες δεν θα τηρούσαν τους ε, κανόνες, κάτι το οποίο ε, δεν ήταν η επίσημη θέση της, Βρετανικής, ε, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ήταν απλά μία πρόταση. Αυτά ο κύριος Χιούζ. Η δήλωση για την ανάπτυξη και την απασχόληση ζητάει ε, έξυπνη δημοσιονομική εξυγίωση, ε, κάποιες μακρονομικές πολιτικές και μια ενεργή στρατηγική απασχόλησης για να υπάρξει κοινωνική συνοχή. Αυτό ζητάει εδώ από την αρχή της κρίσης το κόμμα μου. Ε, Αντί να έχετε όμω έξυπνη προσέγγιση για δημοσιονομική εξυγίανση, έχετε μία χαζή. Ε, το πακέτο των έξι μέτρων έγινε χειρότερο από αυτή τη νέα συνθήκη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τι επενδύσει για την μελλοντική ανάπτυξη, όπω να είναι τα συμπεράσματα. Αν θέλετε να είστε έξυπνοι, μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα. Ε, μπορείτε, ε, όπω λέει το Κοινοβούλιο, να δημιουργήσετε ένα πραγματικό σύστημα ευρωομολόγων. Ε, να μειωθούν τα επιτόκια για το δημόσιο χρέο και να ε, υπάρξει χώρο για νέε επενδύσει το Συμβούλιο θα μπορεί να ε, συμφωνήσει για αυτό το φόρο χρηματοπιστωτικών αλλαγών και να δημιουργηθούν 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό ήταν έξυπνο. Ελπίζουμε ότι η σχέση του Συμβουλίου, η κατάσταση στο Συμβούλιο να αλλάξει, ούτω ώστε να δοθούν πραγματικά έξυπνες ε, απαντήσεις για την κρίση. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπε ο κ. Κάλλαν, ε, υποτίθεται ότι θλίβεται για το γεγονός ότι γίνεται παράνομος ο σοσιαλισμός με αυτή τη συνθήκη. Α, σας ευχαριστώ που λέτε έτσι τόσο ξεκάθαρα την ε, συντηρητική σας θέση. Ευχαριστώ, η κυρία Μπόλς, ευθυνόντας Σάλντε. Thank you, President. Jobs and growth have made it to the top of the agenda. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απασχόληση και η ανάπτυξη είναι το κύριο θέμα. Επίσης το άλλο είναι η κρίση για τους νέους. Αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός έχουμε πάρα πολλούς άνεργους νέους. Δεν πρέπει να ξεχναμε δυο 2-3 εκατομμύρια και πάνω βλέπετε από το τραπεζικό σύστημα μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, άρα κάτι γίνεται ήδη. Το θέμα είναι όμως αυτή η γενιά θα τον αντιμετωπίσει ή θα μεταβιβάσει τα προβλήματα και την ανεργία στους νέους που δεν έχουν ε, απασχόληση, δεν έχουν σπίτι και αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες αυτής της γενιάς. Και εκείνοι που προσπαθούν να κατηγορήσουν την ε, τράπεζα για τα stress test θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ε, λέγεται ότι θα πρέπει να γίνουν, να γίνουν αυτά τα stress test και να υπάρχουν και προστατευτικά τείχη. Και αυτές οι καθαρίσεις για προστατευτικά τείχη και άλλες καθυστερήσεις οδήγησαν στα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέπιν για την αίμα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω πρώτα απ' όλα το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Έχει καθυστερήσει 10 χρόνια ε, υπάρχει νομισματική ένωση χωρίς να υπάρχει μια δημοσιονομική βάση. Αλλά η λύση αυτή δεν λύνει τα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Η Ελλάδα δεν θα ανακάμψει στην Ευρωζώνη. Η Πορτογαλία είναι στο όριο. Η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία άξαν την ανταγωνιστικότητά τους λόγω του ευρώ. Μεταφορές κονδυλίων δεν θα το αντικαταστήσουν αυτό. Ούτε θα κάνουν τα προβλήματα λιγότερο οξυμένα όπως ε, θεωρεί ο κύριος Σαρκοζή. Ο κύριος Σαρκοζή κάθε φορά που βγαίνει προτείνει νέο κείμενο. Τι χρειάζονται ε, υποψήφιοι σοσιαλιστές. Ο κύριος Σαρκοζή γίνεται κάθε μέρα πιο σοσιαλιστής. Τώρα μιλάμε δε για τσάρο προπολογισμού, ε, ο οποίος ήταν ο κύριος Ρεν. Η Φιλανδία είχε ζήσει υπό τον τσάρο, τα ξέρει αυτά. Αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Κύριε Μπαρόζο, Πρέπει να το έχετε αυτό το ιστορικό μάθημα κατά νου. Α, έχει φύγει ο κύριος Μπαρόζο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σόρεν Μπος Όντεργκαρτ για την ΚΟΕ για ένα Ευχαριστώ. Εκφράζω την έκπληξή μου για τα αποτελέσματα αυτής της Συνόδου Κορυφής. Είναι ακατανόητα. Αν υπάρχουν χώρες που έχουν προβλήματα με την οικονομία τους, τους ε, επιβάλλουμε πρόστιμο. Τσακ, λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί δεν το έχει σκεφτεί κανένα έξυπνο πριν. Είναι τόσο απλό, τόσο αποτελεσματικό. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο και να επιλύσουμε και άλλα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, μια χώρα που έχει πάρα πολλού ανέργου. Δεν είναι δύσκολο. Επιβάλλουμε ένα πρόστιμο. Όταν υπάρχουν πολλοί φτωχοί. Πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Να επιβάλλουμε πρόστιμα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όμω δεν θέλησαν να πάνε τόσο μακριά. Δεν τόλμησαν να πάνε τόσο μακριά. Τα εκατομμύρια φτωχών και ανέργων τα δεχόμαστε χωρί να επιβάλλουμε πρόστιμα. Αλλά αν μια χή χώρα αποφασίσει να κάνει μαζικές δημόσιε επενδύσει. δανειζόμενη για να δημιουργήσει πράσινε θέσεις απασχόληση, α πούμε, στα πλαίσια της οικονομίας, ε, αιωλικής ε, ή ηλιακής ενέργειας. Τότε αμέσως πέφτει ο πέλεκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι χαζός και περιορισμένος τρόπος να ασκούμε έτσι οικονομική πολιτική. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το υποδέχτηκαν με μια γενική απεργία οι Βέλγοι εργαζόμενοι. Ελπίζω να επαναληφθεί αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Η κυρία οι τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε σήμερα εδώ μας, δίνει, μας δείχνει ότι ουσιαστικά οδεύουμε σε μια ενιαία Ευρώπη αν στοχεύουμε να γίνουμε η ενωμένη η ευρώπη των ενωμένων κρατών όπως είναι το μοντέλο πούμε των ηνωμένων πολιτειών έχετε δει ποτέ αξιωματούχο από το μίσιγκαν να επιτίθεται στην υπερχρεωμένη καλιφόρνια όπως κάνουν διάφοροι δημόσιοι ευρωπαίοι πολιτικοί ουσιαστικά πιστεύω ότι όλοι μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποσυνθέσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. κριτική σχόλια ανόητες προτάσεις ανοησίες οι οποίες επιβάλλουν πολιτικές σε χώρες οι, οποίοι, οι οποίες έχουν πολίτες. παρακολουθούμε διαδικασίες καταστρατήγησης της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών. παρακολουθούμε διαδικασίες καταστρατήγησης του των νόμων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ως Ελληνίδα αποδέχομαι κάθε επικοδομητική κριτική για ό,τι έκανε και κάνει η χώρα μου. Αλλά έχει στοιχηθεί όμως όλη η Ευρώπη πίσω από τη μικρή Ελλάδα και όλα τα προβλήματα της κρίσης τα έχει η Ελλάδα. Λέτε και οικοδομήσαμε το ευρώ σε μια πολύ σωστή βάση. Εκεί δεν έκανε κανένας λάθος. Όσο υπάρχει πρόβλημα Ελλάδος υπάρχει και πρόβλημα Ευρώπης. Κάνουμε έκκληση σε όλους εσάς Σταματήστε να ασχολείστε με την Ελλάδα. Εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Και μία έκκληση προς τους Γερμανούς συναδέλφους. Ήδη δημιουργείται χάσμα και έχει όνομα και πρόσωπο και είναι η Γερμανία. Ήδη τα, νο... τα ΜΜΕ στην Νότια Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα λεπτό, αποκαλούν τη Γερμανία ο έφηβος ηγεμόν. Προβληματίζομαι και φοβάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε μια πλάτη να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε παρότι δεν είχα χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε λοιπόν την ε, νέα σύνοδο η οποία για το κόμμα στο ΠΒΒ ήταν τελείως άξιτη, δεν αποφασίστηκε τίποτα. Απλά ελπίζουμε για το καλύτερο και όλα θα πάνε καλά και με την Ελλάδα και με την ανεργία των ε, ένων. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν εγκαταλείπει η Ελλάδα την νομισματική ένωση και το κούρεμα το 70% δεν θα ωφελήσει τίποτα. Και εγώ το ξέρω και εσείς το ξέρετε και όλοι οι ανεξάρτητοι οικονομολόγοι το ξέρουν. Παίζουμε εδώ πέρα με τα λεφτά των ε, φορολογουμένων πόκερ και η δημοσιονομική πειθαρχία η οποία φαίνεται πως είναι η μαγική λέξη του 2012. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς μπορείτε εσείς κύριε Μπαρόσο να λέτε πως ε, θα πρέπει να μειωθούν ακόμα και οι ε, μικροί πορτογαλικοί μισθοί και επιδόματα. Δεν τα πιστεύει αυτά βλέπετε και η αγορά. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Φοβάμαι πως ρίχνουμε λάδι στην ε, φωτιά. Αυτή τη στιγμή στη Νότια Ευρώπη οι μισοί νέοι μέχρι 25 ετών είναι άνεργοι. Και αντί να δημιουργήσει ε, ευημερία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξελιχθεί σε έναν εφιάλτη. Και τι βλέπουμε στο νέο αυτό κείμενο το οποίο εγκρίθηκε, θα χρειάζεται να περιμένουμε να εγκριθεί και να τεθεί ενισχύ. Δεν ξέρω αν έχουμε αυτή την ε, πολυτέλεια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόιλ, ο οποίος είναι ο νέος επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας της σου συγχαρητήρια. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερα λύση, αλλά νομίζω ότι αυτή η λύση ήταν καλή. Πολλέ φορέ στην πολιτική υπάρχουν καταστάσει στις οποίες θα πρέπει να επιτύχει κανένα το κατοδυνατόν καλό, να ικανοποιηθεί και να προχωρήσει μετά βήμα προ βήμα. Αυτό που είτε επιτευχθεί είναι φυλασμιόν με αυτό που αποφασίσαμε πριν από 6 μήνε μέσα στα πλαίσια του Six Pack. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι γίνεται. Θελήσαμε να ή ακολουθήσουμε μια πολιτική λιτότητας, να μειώσουμε τα χρέη, να προωθήσουμε μια πολιτική ανάπτυξη. Δεν γίνεται τώρα αυτό ακριβώς όπως το θέλαμε, είναι σωστό. Οι συνάδελφοι συμμετείχαν εκεί και προσπάθησαν να βελτιώσουν κατά το δυνατόν το αποτέλεσμα. Το είπε ο Έλμαρ. Και τώρα βλέπουμε εδώ τους προέδρους των μεγάλων πολιτικών ομάδων που ακολουθούν μια πολιτική κομματική της χειρής της μορφής όταν έχουμε τέτοια προβλήματα στην Ευρώπη να υπάρχει αυτό το θέαμα εδώ είναι απαράδεκτο. Σοκάρομαι, σοκάρομαι κυριολεκτικά. Όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, κύριε Πρόεδρε, δεν επιτρέπεται να ακολουθεί τέτοια φτυχνή κομματική πολιτική. Δηλαδή δεν πρέπει να προωθούμε την ενότητα της Ευρώπης και εμείς να προωθούμε αυτή την ε, την διάσπαση. Αν χρησιμοποιήσει κανένα τέτοια λόγια όπω πολλοί πρόεδροι πολιτικών ομάδων, θα πρέπει να ντρέπεται. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οι μεν του 10 αυτόν τον τρόπο και δεν θα πετύχουμε ποτέ έτσι μια ενωμένη Ευρώπη. Πρόεδρε, θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Η συνάδελφο κυρία Χάρμ θέλει να σα υποβάλει μια ερώτηση. Ε, το φανταζόμουν, ναι. Εάν κατάλαβα σωστά, τότε αυτό το six-pack, το δέσμευτη των 6 μέτρων, που αποφάσισε εδώ πλειοψηφικά το σώμα, είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που λειτουργεί ήδη και ε, η οικονομική ένωση από πότε θα αρχίσει να λειτουργεί και σε ποιες χώρες θα οδηγήσει σταθερότητα. Από πότε θα λειτουργήσει και ρορόιλ. Μα δεν μπορώ να σας δώσω καμία ημερομηνία, αλλά γρήγορα, γρήγορα το ξέρετε. Και ξέρετε και ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς χρειάζονται μία προθεσμία εφαρμογής και εσείς επικρίνετε όχι τις ε, προθεσμίες αλλά το περιεχόμενο, τη διαδικασία αυτών που αποφασίστηκαν το, τη Δευτέρα. Απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Η κυρία Τράουπεν έχει το λόγο. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θέλω να αρχίσω να κάνω μικροπολιτική κυρία Ρόλη, σας διαβεβαιώ. Γιατί νομίζω ότι αυτή η συνθήκη μας ε, κάνει τσεκμάτα μάτα και λυπάμαι γι' αυτό. Ε, λυπάμαι για την αποτελεσματική. Για να απαντήσουμε στις αγορές απέναντι στην κρίση, γιατί δεν αποκαθιστά την εμπιστοσύνη. Βλέπουμε τα προβλήματα της Πορτογαλίας, της Ελλάδας. Βλέπουμε δύο χώρες που είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες, η Γαλλία και η Γερμανία, να μειώνουν στο ίμιση το ποσοστό ανάπτυξής τους. Υποτίθεται ότι όλα αυτά θα έπρεπε, να, θα έπρεπε αυτή η συνθήκη, ας πούμε, να ρυθμίσει τα πράγματα. Θα έπρεπε η ΕΚΤ ε, με την ρευστότητα που έχει στις τράπεζες να μας βοηθήσει να φύγουμε από την κρίση. Εδώ οι εκλογείς μας μας έστειλαν εδώ πέρα για να βρούμε λύση. Είναι οι άνεργοι, είναι οι νέοι που θέλουν να έχουν προοπτική, θέλουν, ε, είναι οι συνταξιούχοι. Δεν μπορούμε να επικρίνουμε απλώς μια συνθήκη που ε, είναι βασισμένη μόνο στη δημοσιονομική πειθαρχία και που ε, δημιουργεί ε, μια κάστα που εποπτεύει απλώς τους άλλους, θα πρέπει να επαναστατήσουμε ενάντια σε αυτά τα αποτελέσματα και να κάνουμε προτάσεις. Εγώ έχω προτάσεις, δεν θέλω απλώς να καταδικάσω. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να προτείνουμε σήμερα για την Ευρώπη είναι ένα σύμφωνο ευρωπαϊκό ευθύνη ε, διακυβέρνησης διακυβέρνηση και ανάπτυξη. Θα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτούμε αυτή τη συνθήκη, ούτω ώστε να υπάρχει ένα πραγματικό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με βιομηχανική πολιτική για να δουλέψουν τα εργοστάσια μα και οι εργαζόμενοι στον τομέα τη ενέργεια και του περιβάλλοντο. Να υπάρξουν ευρωομόλογα. Ε, τα ξεχάσαμε δυστυχώ, τα διαγράψαμε να υπάρξει και δημοσιονομική ρύθμιση, υπάρχει πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη. Αυτά πρέπει να προωθήσουμε στο κοινοβούλιο μας. Μάουρο, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο υπερασπιστήκατε όχι μόνο τα πλεονεκτήματα της ε, ε, συνέλευσής μας, αλλά και τη δημοκρατικότητα της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο ε, την καλή δουλειά που έκανα ο κύριος Μπρόκ, ο κύριος Φερχώστα και ο κύριος Γκουαλτιέρη. Έχουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε τι προτάσει που θα κάνει. Μιλάνε για τι προτάσει που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. καινοτομήστε. Ε, ανανεώστε την διαδικασία λήψη των αποφάσεων Και εκ των προτέρων να λάβετε υπόψη σα ε, τις ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων, όχι εκ των υστέρων. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σήμερα ακούσατε του κουφού και τυφλού εθνικιστέ που ξεχνούν τα 65 χρόνια ειρήνης της Ευρώπης ε, και θεωρούν, και θεωρούν ότι αυτό ήταν, το είχαμε από πάντα. Ξεχνούν ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνα τη Ευρώπης. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί ε, αρχηγοί δεν ξέρουν πού να στρέψουν την κεφαλή τους, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ένα μισή λεπτό. Θέλω να σχολιάσω τα συμπεράσματα του, της Σύνοδου Κορυφής. Είπαμε ότι το Κοινοβούλιο δούλεψε για να περιορίσει τις ζημιές αυτής της ε, επιλογής που δεν ήταν και η καλύτερη. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο σε αυτή τη δύσκολη διαπραγμάτευση είχε αυτή την ε, θέση και βοήθησε ούτως ώστε να αποφύγουμε το χειρότερο. Υπήρχε ο κίνδυνος η νέα συνθήκη να υποσκάψει το δίκαιο το ευρωπαϊκό, να βάλει μηχανισμούς και διαδικασίες εξωτερικούς από την Ένωση και σε αντίφαση με, τους, με, το, την εθνική νομοθεσία. Το, ξεφύγαμε από αυτόν τον κίνδυνο. Το Κοινοβούλιο Κομισιόν ε, απέτρεψε αυτόν τον κίνδυνο. Τώρα θα πρέπει η νέα συνθήκη να εφαρμοστεί μέσα από την ε, ενωσιακή νομοθεσία. Ε, οι παράμετροι για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους ε, άλλαξαν ε, και εντάχθηκαν στο σημερινό ε, πλαίσιο και δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ορίζοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Παρ' όλα αυτά, λείπουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι απαράδεκτα. Όπως, παραδείγματος χάρη, η μειωμένη παρουσία του Κοινοβουλίου στη Συνόδου Κορυφής μόνο αν οι προτάσεις που θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, ε, ο φόρος για τις δημοσιονομικές αλλαγές, ε, τα ομόλογα σταθερότητας, ε, τα ομόλογα έργων, μόνο αν αυτά τα δεχτούμε η Ευρώπη θα μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση, γιατί αλλιώς θα, η κρίση μπορεί να εμβαθυνθεί λόγω αυτής της δημοσιονομικής μονομερούς λιτότητας. Ευχαριστώ κύριε Κολτιέρη και σας ευχαριστώ επίσης και για την διαπραγμάτευση και τον κύριο Φερχόφστατ και τον κύριο Μπρόκ. Εντάξει, σας σας ξέχασα γιατί είστε και πρόεδρος ομάδας, αλλά νομίζω πως εκπροσωπήσατε εξαιρετικά το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Λεγκρίπ για το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να Πλησιάσω την γαλλική πτυχή του ΕΛΚ όσον αφορά την οικονομική διαδίκηση και την υποστήριξη για τα βασικά συμπεράσματα στο οποίο κατέληξε το Συμβούλιο. Να μην ξεχνάμε, αυτή η συνθήκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για περισσότερη ολοκληρώση οικονομική, δημοσιονομική και περισσότερη οικονομική σταθερότητα. Το ξαναπούμε. Δεν μπορεί να ξανυπάρξει μόνιμη ανάπτυξη ε, και απασχόληση χωρίς να εξηγιαθούν τα δημόσια οικονομικά δεν είναι μια συνθήκη εκείνη η οποία θα μπορέσει να ξαναδώσει ζωή στην ανάπτυξη, αλλά μια συνθήκη που οδηγεί σε αμοιβαία δέσμευση μπορεί να οδηγήσει σε ευθύνη και υπευθυνότητα, όπως ε, μια που ο πρόεδρος ε, της ε, Σοσιαλικής Ομάδας εισήγηγε μια πολιτική, αν θέλετε, πτυχή στη συζήτησή μας, αναφέρομαι στις προεδρικές εκλογέ στη Γαλλία. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς στο ΕΡΚ θεωρούμε απολύτως ανεύθυνες οι δηλώσεις του σοσιαλιστή υποψήφιου ότι θέλει να ξαναδιαπραγματευτεί τη συνθήκη που υπάρχει. Γιατί, με ποιον και πώς. Είναι τελείως ανεύθυνα αυτά που είπε. Δεν είναι μια δήλωση που σέβεται τις υποχρεώσεις της γαλλικής, ε, του γαλλικού κράτους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούλμαν ε, που εξελέγει ε, επικεφαλής της ε, αντιπροσωπεία στη σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δούμε τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα, την ημέρα της ε, Συνόδου οι αγορές ε, αξιολόγησαν τα δεκαετή ομόλογα της Πορτογαλίας με 17% για τα δε πενταετή με 20%. Αυτά για το κατά πόσον καθυσίχασε τις αγορές η σύνοδος αυτή και για το τι σημαίνει ε, για τις αγορές η νέα αυτή η διακυβερνητική συνθήκη. Και αν αναρωτιέται κανείς από πού προκύπτει αυτή η ανησυχία, ίσως από τα οικονομικά δεδομένα και από την αίσθηση πως δεν επαρκούν αυτά τα οποία έχουν γίνει. Κύριε Πρόεδρε Σούλτς, θα ήθελα να πω πως το θάρρος και η σαφήνεια με την οποία μιλήσατε εσείς εξ ονόματος Κοινοβουλίου και λέτε ναι, θα υπερασπίσουμε την κοινοτική μέθοδο, ναι, πρέπει να κάνουμε οικονομία αλλά και επενδύσεις για να μπορούν να ανθίσουν οι οικονομίες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά τα οποία είπατε και νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό για να τυχθεί περαιτέρω η κοινωτική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σάριος Βόλσκι για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να αναφέρω μία προσθέμενη αξία που θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε ε, όσον αφορά την εφαρμογή του πακέτου αυτού. Αντιμετωπίζουμε ένα τεστ αξιοπιστία τη πολιτική μα από τι χρηματαγορέ. Πρέπει να δράσουμε σε ένα πνεύμα ενότητα και αλληλεγγύη και να μην έχουμε άσκοπε διαιρέσει. Όσοι είναι πιο υγιεί μακροοικονομικά θα πρέπει να διευκολύνουν αυτού που είναι λιγότερο. Αυτό με οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει ένα μοίρασμα του χρέους, αυτό είναι μια προσθέμενη αξία, με αντάλλαγμα βεβαίως μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά το έλμα δεύτερον, δεδομένη του ότι 12 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης ε, ξεπερνάνε το χρυσό κανόνα του λόγου χρέος προς ε, ΑΕΠ, ενώ 8 μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν, από τα 8, τα 7 δεν το τηρούν, μπορούμε να πούμε πως αυτή την ε, στιγμή πριμοδοτούν τα μη κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τα νυν κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Έχουμε άρα μία προσθέμενη αξία της Ευρωζώνης και είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να ε, δεχτεί αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει κυρία Φερέιρα τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Αυτή η συνθήκη είναι περιττή και ανώφελη και επιπλέον επικίνδυνη. Καταρχάς γιατί θα ενισχύσει με άκαμπτους κανόνες και με τιμωρίες ένα φάρμακο το οποίο δεν λειτουργεί. Ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό ο οποίος δεν διαφοροποιεί ανάμεσα στην ανορεξία και στην αρρώστια και που συζητάει μαζί με τον ασθενή ε, το πιθανό του θάνατο. Πόσε χώρε πρέπει να αρρωστήσουν για να καταλάβει το Συμβούλιο ότι η διάγνωση είναι λάθο. Έχουμε 23 εκατομμύρια ανέργους, 6 εκατομμύρια νέων ε, δεν έχουν καμία ελπίδα να βρουν δουλειά. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν κατάλαβαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, δεν γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα. Και το να μην ε, προσαρμόζουμε τα μέσα, τα, το φάρμακο στην αρρώστια είναι αυτισμός. Ίσως κάνετε ιδεολογικές ε, επιλογές, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Υπάρχει μια άλλη ατζέντα που η άλλη ατζέντα δεν βασίζεται σε λόγια αλλά σε πράξεις. Παραδείγματο χάρη τα ομόλογα έλγων, η ενίσχυση των προϋπολογισμών χάρη σε ένα φόρο των κερδοσκοπικών συναλλαγών. Θα πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τις χώρες από υπερβολικά και καταχρηστικά επιτόκια. Χρειαζόμαστε δράσεις και όχι λόγια. Η κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. μετά από τέσσερα χρόνια από την έναρξη της κρίσης δεν υπάρχει ακόμα μια σταθερή απόφαση για έξοδο από αυτή όλης της ευρώπης. το σύμφωνο σταθερότητας γνωρίζουμε όλοι ότι δεν ήταν πραγματικά αναγκαίο σε νομικό επίπεδο προφανώς ήταν αναγκαίο μάθημα πειθαρχίας ή και απειλής για αυτούς που παρεκκλίνουν από τους κανόνες Ας δεχθούμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια λύση, αφού όλες οι άλλες δυνατές είναι χειρότερες για τα ισχυρά κράτη-μέλη της Ένωσης. Η ύφεση, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται από μόνη της να δώσει απάντηση στο πρόβλημα σε καμιά χώρα, ιδιαίτερα στη δική μου. Η δημοσιονομική πειθαρχία και το πρόγραμμα λιτότητος είναι απολύτως αναγκαία αλλά χωρίς ανάπτυξη αποτελούν απλώς μια αδιέξοδη πολιτική με ολέθρια αποτελέσματα όχι μόνο για τις χώρες που εφαρμόζεται αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. κύριε Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι που μεταξύ των βασικών θεμάτων της Συνόδου Κορυφής ήταν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αλλά από το Δεκέμβριο και μετά βλέπουμε ότι παίρνονται αποφάσεις χωρίς να βελτιώνεται η κατάσταση. Παίρνονται αποφάσεις διακυβερνητικές οι οποίες ε, δεν είναι πάντα αναγκαίες. Η τελευταία δεν ήταν αναγκαία. Επίσης αυτή η νέα συνθήκη ουσιαστικά δεν πάει και πολύ πέρα από το six pack. Εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Λυπάμαι μάλιστα που ούτως ή άλλως στο παρελθόν ε, με το six pack δεν πετύχαμε τίποτα και πήραμε αποφάσεις ε, που μας ανάγκασαν να βουλιάξουμε ακόμα πιο βαθιά. Χρειαζόμαστε έργα και όχι λόγια. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη. Δεν νομίζω ότι με αυτή τη συνοκορυφή κάναμε ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός. Εξάλλου δεν υπέγραψαν όλοι αυτή τη νέα συνθήκη. Πάντως πιστεύω ότι μέχρι το Μάρτιο έχουμε χρόνο για να καλύψουμε τα κενά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε δει μέχρι στιγμής να υπάρχουν. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Eye, όπου θα ακουστούν όσοι ε, ζητάν ε, το λόγο αυθορμήτω. Βεβαίω εδώ και μια μισή ώρα μιλάνε οι συνάδελφοι αυθορμήτω. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε με τον κύριο Λούχαν, ο οποίος είχε ζητήσει το λόγο στην αρχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όσον αφορά την ανεργία των νέων, θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο. Η δε κατάσταση για τους ε, νέους ε, βελτιώνεται με ποια έννοια, με την έννοια ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν αφορούν κυρίως τους νέους. Θεωρώ πως ε, ένας βασικός τρόπος επίτευξης ε, των στόχων αυτών είναι η πολιτική συνοχή. Σε αυτή τη στιγμή, σε εθνικό επίπεδο, ε, βρισκόμαστε στην φάση του προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020. Κομισιόν και Συμβούλιο θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος ε, στην απασχόληση των νέων και να στηρίξουν προγράμματα με επαρκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ποδηματά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω ασφαλώς ότι δεν συμμερίζεστε ορισμένες από τις ακραίες και προσβλητικές αναφορές που έγιναν από ορισμένους μονίμως φωνασκούνται σε αυτή την αίθουσα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα ούτε να απευθυνθώ σε αυτούς ούτε να σχολιάσω τα λεγόμενά τους. Θέλω όμως να απευθυνθώ στους υπόλοιπους συναδέλφους ε, και να τους ζητήσω να αναλογιστούμε πού οδηγούν τα στερεότυπα οι ισοπεδωτικές αντιλήψεις και οι αναφορές απέναντι σε μια χώρα και σε έναν ολόκληρο λαό που δοκιμάζεται σκληρά από την κρίση και θέλω να επισημάνω έχει φύγει ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Μπρόκ ότι δεν αμφισβητώ τις προθέσεις της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων εδώ. Όμως όταν είμαστε ειλικρινείς ότι θέλουμε να βοηθήσουμε μια χώρα να ολοκληρώσει την προσπάθειά της δεν θα πρέπει να την προσβάλλουμε διότι όπως είπε και ένας άλλος γερμανός ο Σίγμουρ Γκάμπριελ όταν βάζει ένα λαό να διαλέξει ανάμεσα στην εθνική αξιοπρέπεια και την βοήθεια είναι σαν να αγνοείς βασικά διδάγματα της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να πω πως πρώτα απ' όλα θεωρώ πως ως έναν βαθμό σερνόμαστε από τον ένα κανονισμό στον άλλον και ήταν δύσκολο να μπορούμε να έχουμε μία αντίληψη των γεγονότων χωρίς τα θεσμικά μας όργανα. Ο κύριος Δράγκη είπε πριν από δύο εβδομάδες είπαμε πως μπορούμε να έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ε, ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομική πειθαρχία. Συμφωνώ, ναι, αλλά μεγαλύτερη έμφαση παρακαλώ στην ανάπτυξη. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένας νέος ορισμός του τι ή θεωρείται η οικονομία της αγοράς. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου θεωρώ πως ο ιδιωτικός τομέας ρυθμίζει τον δημόσιο και δεν υπάρχει καμία λογοδοσία. Οι ολιγάρχες κυβερνούν ορισμένα τμήματα των αγορών. Λίγη περισσότερη προσοχή στο τι κάνουν οι αγορές στον δημόσιο τομέα και σε όλα τα κοινοβούλια και κυβερνήσει. Και ας προσπαθήσουμε εμείς να έχουμε ηγετικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι κι εγώ, όπως πολλοί συνάδελφοι, έτσι και εγώ είμαι κάπως διχασμένοι. Από τη μία συμφωνώ με τους Ευρωπαίους ηγέτες που λένε πως χρειάζεται άμεση δράση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική. Από την άλλη είμαι πεπισμένη πως η αφετηρία μας δεν είναι η σωστή. Ναι, δεν μπορούμε χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα και αυστηρού κανόνες, αλλά κατά την άποψή μου η ρίζα του προβλήματος ήταν πως δεν έχει δοθεί αρκετή βάση στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Κατανοητό βεβαίω οι περισσότεροι ηγέτε ασχολούνται με μέτρα λιτότητα. Μέγα λάθος Επιπλέον δεν είμαι σίγουρη για την μορφή αντιμετώπιση της κρίση. Πρέπει να ακολουθήσουμε την κοινωνική μέθοδο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ευρώπη να απομακρυνθεί από αυτά τα οποία εκπροσωπεί. Η Ευρώπη συνεργάζεται ανεξαρτήτω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Πέρα από αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο είναι άμεσα ερετό. Ο πρόεδρος μας λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, βλέπω τώρα την κυρία Ματίας εδώ πέρα που έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Μπαρόζος, τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανε μια παρουσίαση PowerPoint, πολύ διδακτικό, με γραφικές παραστάσεις, ε, για τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης ε, που έγινε ε, για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες. Έχω φρίξει, γιατί το βάρος των εργαζομένων ήταν ο πέμπτος τροχός της αμάξης Ε, και το πέμπτο μέλημα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή η ύφεση, ε, η έλλειψη πίστοσης, κονδυλίων δηλαδή, οι συνθήκες, της, οι επιπτώσεις της κρίσης. Κάτι μου διαφεύγει. Κύριε Φανρόμπουη, γιατί οι κυβερνήσεις ασχολούνται μόνο και προωθούν μόνο τη λιτότητα. Γιατί επιμένετε στη μείωση των μισθών ως μόνη λύση. Τι δεν έγινε σωστά. Ε, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι σωστές οι ερωτήσεις που θέσατε δεν είναι σωστές. Είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσει, μου, σας παρακαλώ, κύριε Φανρόμπουη. Πέρα από τις ε, λέξεις, πέρα από τα λόγια. Ο πρόεδρος διακόπτει όμως την ομιλήτρια. Έχω άλλους δύο συναδέλφους και μπορώ να τους δώσω το λόγο και μετά τελειώνουμε οριστικά. Ο κ. Ποτασίεβιτς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση καθώς και η συζήτηση στον Ευρωπαϊκό Τύπο καταδείκτουν ότι δεν έχουν πληρωθεί όλες οι προσδοκίες ε, από την διάσκεψη κορυφής της Δευτέρας. Είναι αλήθεια αυτό από την άλλη μεριά όμως ήταν ε, μία διάσκεψη κορυφής ε, με καλές και σοφ... καλούς και σοφούς ε, συμβασμούς. Υπάρχει περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία και καλύτερες προοπτικές για τις οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης και μπορέσαμε επίσης να αποτρέψουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων με διαφορετικά θεσμικά όργανα πολωνική κυβέρνηση ξεκίνησε διπλωματική επίθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σόλτς που προώθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε αυτές τις δυσαρέσκειες για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και δεν θα είναι ούτε αυτή τη φορά η τελευταία. Καταρχάς, είναι μονομερή τα συμπεράσματα. Ασχολούνται μόνο με τα ελλείμματα. Και ως φάρμακο ε, μιλάνε για το σεβασμό κάποιων στόχων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοσιονομική ένωση. Ε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που προωθούμε είναι ε, μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας με επιβολή προστήμων. Το κοινοβούλιο μας τι θέλει. Θέλει να... Δεν έχει καταλάβει ότι χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση για να βγούμε από αυτή την κρίση. Ε, αν δεν κάνουμε κάτι, κάτι θετικό, ε, δεν υπάρχει περίπτωση ο ασθενής να αναρρώσει. Ευχαριστώ. Ε, Πρωτού να δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο και στον κύριο Φανλομπόη, έχω να σας πω κάτι. Αυτό το catch the eye εισήχθη και παρακαλώ να το σκεφτούν αυτό οι πρόεδροι πολιτικών ομάδων. Εισήχθη, λέω, ότι ώστε αυθόρμητα στη συζήτηση, στο τέλο τη συζήτηση, να δίνουμε το λόγο στου συναδέλφου. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ότι το catch the eye είναι κατά κάποιο τρόπο ένα δεύτερο κατάλογο των αγορετών. Όπου τίθεται υποποίηση να δώσει το λόγο σε κάποιου συγκεκριμένου. Δεν το κάνω αυτό. Εγώ προσανατολίζουμε στην νοθαρμισμό των συναδέλφων και σας παρακαλώ στο μέλλον, στο τέλος της συζήτηση, να μπορούμε αυτά να δίνουμε το λόγο σε εκείνους που είναι παρόντες και ζητούν το λόγο. Αλλιώ είναι άδικη η διαδικασία. Ο κ. Σεύκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ για την πολύ έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τι νέε ιδέε που ακούστηκαν σε αυτή τη συζήτηση γιατί δείχνεται το πραγματικό συνέστημα που υπάρχει στον κόσμο ότι αυτή η συνοσκορυφή ήταν πολύ κρίσιμη. Σε αυτή την χρονική στιγμή η βασική εστίαση είναι στην ανάπτυξη και αυτό ήταν σημαντικό που υπόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών μας είναι η ανάπτυξη και είναι η απασχόληση. Φυσικά υπήρχαν και πολύ σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν για να υπάρξει πιο ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους διαπραγματευτές, τον κύριο Φερχόφστατ, τον κύριο Γκουαλτιέρη και τον κύριο Μπροκ για τη θαυμάσια δουλειά και την καλή συνεργασία που είχαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επανέρχομαι τώρα στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Νομίζω ότι οι συζητήσεις για την ανάπτυξη και ο κύριος Φερχόφστα θα μιλήσει για τη θετική στάση και τη σημασία που δώσαμε στην ανάπτυξη, ήταν πολύ σημαντική. Δεν συμφωνώ με αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης διαλύοντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ήδη στο 18ο και 19ο αιώνα το είχαμε στην Ευρώπη. Ας μην οπισθοχωρήσουμε για την εστίαση που υπήρχε, υπήρξε στη νεότητα. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να βοηθήσουμε τους νέους, τη νέα γενιά, ούτω ώστε οι 7,5 εκατομμύρια νέοι που δεν απασχολούνται, που δεν πάνε σχολείο ή πανεπιστήμιο, να απασχοληθούν, ε, είναι πολύ σημαντικό. Η επιστολή στα 8 κράτη-μέλη εστάλει και το Φεβρουάριο η κοινή δράση θα δρομολογήσει και θα κινητοποιήσει τα νέα κονδύλια αυτά υπέρ της απασχόλησης των νέων. Θέλουμε την συνεργασία σας ε, και την υποστήριξή σας σε αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη. Στο σημαντικό θέμα της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Από τη συζήτηση που κάνατε και από τη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκύπτει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εξυγίαση χωρί ανάπτυξη. Το τελευταίο χρόνο ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη σωτηρία του ευρώ. Προσπαθούμε να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Τώρα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει μια κάποια ε, σταθεροποίηση. Μπορούμε να ασχοληθούμε με την ε, ανάπτυξη, κάτι που θα βοηθήσει πολλέ οικογένειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί και άκουσα τη συζήτηση που έγινε, ορισμένοι Μίλησα, βέβαια με πολύ ε, ζωφερότερα λόγια για τη συνοκορυφή από ό,τι πρέπει. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο διατήρησαν την, κοινωνική, την κοινοτική μέθοδο. Και με, είναι σίγουρο ότι η εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην οικονομική διακυβέρνηση είναι εξασφαλισμένη. Και αυτή η συνθήκη τελικά μέσα σε πέντε χρόνια θα ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά πράγματα, είναι ωφέλη και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε θετικά και όχι με ζωφερό μάτι και πνεύμα. Τώρα, συμφωνώ με τον κύριο Ντάουλ σε ό,τι αφορά την ε, σημασία της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας θα αυξήσει το ε, εμπόριο κατά 41% σε αυτές τις υπηρεσίες. Θα αυξηθούν κατά 21% οι άμεσες ξένες επενδύσεις. θα έχουμε από μισό μέχρι 1,5% αύξηση του ΑΕΠ. Πού αλλού μπορούμε να βρούμε τέτοια εύκολη, τέτοιο, τέτοιο εύκολο δυναμικό ανάπτυξης. Είναι κρίμα που παρόλα τετοιο ευκολο δυναμικο αναπτυξης ειναι αυτή η οδηγία ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Και θα ξεκινήσουμε τι διαδικασίε επί παραβάση εναντίον των δύο κρατών μελών που δεν την έχουν εφαρμόσει σωστά. Ο κύριο ε, Φερχόφστα τον έφερε τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Σα διαβεβαιώ ότι τονίστηκε και από μένα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και από τον πρόεδρο της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι όταν θα έχουμε την ε, ευκαιρία να μειώσουμε το κόστος κατά 80% θα πρέπει να προχωρήσουμε, να αρπάξουμε την ευκαιρία. Και χαίρομαι λοιπόν ότι τώρα έχουμε τουλάχιστον την προθεσμία και μέχρι τότε θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Μιλάμε για τον Ιούνιο του μέχρι τον Ιούνιο, όπου θα γίνει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και είναι κρίμα που οι τρει χώρε αυτέ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για να βρούμε λύση για το πού θα εδρεύει ο νέο οργανισμό, η νέα υπηρεσία. Τώρα, κύριε Σφόμποντα, για τα σχόλιά σα για το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και, και κύριε Φερχόφστατ, ε, για τα σχόλιά σα για τα ευρωομόλογα. Ο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι σημαντική πρόταση αυτή. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Κάναμε μια δύσκολη πολιτική συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν ε, οδήγησε αποτελέσματα, αλλά δεν παρετηθήκαμε και ούτε παρετιόμαστε μετά από κάθε δύσκολη πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο. Γιατί έκαναμε έτσι, δεν θα υπήρχε κανένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Ε, θα συνεχίσουμε και θέλουμε την υποστήριξή σα. Και πιστεύουμε ότι στο τέλο όλα τα κρατη θα υπάρξει. συνειδητοποιήσουν ότι είναι χρήσιμο αυτό το μέτρο. Και ότι θα υπάρξει επιμερισμό του βάρου. Ε, και ότι θα υπάρξει ένα υγιές ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω στα ορθολογικά επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα υπέρ αυτού του φόρου είναι πολύ ε, ορθολογικά. Πιστεύω ότι τελικά θα ε, επικρατήσουν. Τα ευρωομόλογα και τα ομόλογα σταθερότητα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι θαυμάσει σταθεροποιητικοί και επενδυτικοί μηχανισμοί. το δείξαμε ξεκάθαρα στο εγγραφό μα με τι διάφορε επιλογέ που έχουμε. Τώρα συνεχίζει τη συζήτηση. Είναι δύσκολη συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι οι νέε προσπάθειες για την ε, δημοσιονομική εξυγίανση αυξάνουν την εμπιστοσύνη των κρατών μελών και την εμπιστοσύνη που έχουν τα μέσα στα ΔΕ σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που έχουμε για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών μας. Πιστεύω ότι θα έρθει η μέρα όπου θα χρησιμοποιήσουμε τα ευρωμόλογα, τα ομόλογα σταθερότητας και θα είναι πολύ, σημαντικά, ε, πολύ σημαντικοί μηχανισμοί σταθεροποίησης και επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν πρόβλημα, όπως είπε ο κ. Φερχόφστατ. Μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό χρηματοδότησης από 75% ε, σε 85% για την Ελληνία, την Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία. Τώρα, ε, για την Ελλάδα μπορούμε να το αυξήσουμε το ποσοστό αυτό από το 75% στο 95%. Ε, θα βοηθήσουμε επίσης και τις ελληνικές αρχές για να απορροφήσουν καλύτερα τα κονδύλια που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτ. Στον λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κύριε Φαντρόμπα. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως το είπα και εισαγωγικά, η πολιτική της ανάπτυξης και απασχολής είναι πολιτική σε διάφορα επίπεδα. Βράχει πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, οικονομική πτυχή, η συγκεκριμένη πτυχή της πολιτικής απασχόλησης, το τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο των κρατών μελών και το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ένωσης. Βραχυπρόθεσμα τώρα καταρχήν και ελπίζω να είμαι σύντομα συνολικά. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι βρισκόμαστε τώρα σε μία περίοδο ύφεσης αλλά ότι ερχόμαστε από δύο χρόνια θετικής ανάπτυξης της τάξη του 2% στην ε, Ευρωζώνη και μέσα σε όλη την Ένωση. Η περίοδος που έχουμε πίσω μας λένε πολλοί ότι είναι μια ε, περίοδος ύφεσης. Όχι, όχι δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν ε, βέβαια εκείνες οι χώρες που βρίσκονται υπό την πίεση των αγορών και όταν κοιτάξω όμως το μέσο όρο το 2010, το 2011 ήταν χώρες ε, με ανάπτυξη και απασχόληση και μάλιστα σε μια χώρα που γνωρίζω καλύτερα από άλλες. Το Βέλγιο το 2010 και 2011 δημιουργήθηκαν 100.000 θέσεις απασχόλησης. και 7.000 το 2009 σε μια ε, χρονιά κρίσης και το 2012 ακόμα θα υπάρχει θετική εξέλιξη. Υπάρχουν προβλήματα σε πολλές χώρες και σε πολλές ε, περιφέρειες. Αλλά ήθελα να σας τονίσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη αυτά για το πρόθεσμο; ήταν. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και συμφωνούμε πάνω σε αυτά είναι να υπάρχει μια εμπιστοσύνη στη ζώνη ευρώ. Όταν επανέλθει η εμπιστοσύνη στη ζώνη ευρώ οι καταναλωτές και επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτό θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Το είδαμε το 2009 ότι όταν επανήλθε η εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη τράπεζες υπήρξε εκ νέου οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτά να εργαστούμε. Επίση, η ενεργεία δεν είναι τόσο καταστροφική όπως λέγεται. Ή τα spread. Τα spread σχετικά με τη Γερμανία μειώθηκαν σημαντικά για την Ιταλία και την Ισπανία. 1,6 για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο του spread που πριν, λίγο, πριν από καιρό. Δεν σας λέω ότι φτάσαμε στο στόχο, αλλά σας λέμε ότι υπάρχει μια επαναστροφή θετική και δεν θα αναφέρω στην Ελλανδία, όπου υπάρχει μείωση σε σχέση με το ΔΟΜΠΟ της τάξης του 7%. Τώρα, αρκεί αυτό? Όχι. Βρίσκομαι στο, σημείο στροφής? Ναι. Και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Βραχυπρόθεσμα. Η λύση δεν είναι να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα και να αυξηθούν τα ελλείμματα. Δεν είναι αυτή η λύση. Την προσπαθήσαμε. Απέτυχε. Ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοί που άρχισαν την ίδια πολιτική δημοσιονομικών ε, κινήτρων θα, ε, πρέπει να επανέλθουν σε πιο ορθόδοξη πολιτική. Εκτός αυτού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πολλές φορές ένα έλλειμμα ανοιχτό μεν αλλά διαρθρωτικό. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια λεγμών θα πρέπει να δούμε σε κάθε περίπτωση τι γίνεται. Δεν είναι το 0,5 έλλειμμα κάθε στιγμή. Θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση και υπάρχει να δούμε αυτή την ε, δομή. Βραχυπρόθεσμα. Κάθε μειονέκτημα έχει πλεονέκτημα. Η μείωση της ε, ισοτιμίας του ευρώ βοηθάει τις εξαγωγές μας. Τώρα, βραχυπρόθεσμα, υπάρχουμε στρατηγική του 2020 την κοροϊδεύουμε, τη συγκρίνουμε με τις στρατηγικές Λισαβόνες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ενσωματώσαμε τη στρατηγική του 2020 στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στο Six Pack το λεγόμενο. Από πλευρά λοιπόν και του Κοινοβουλίου υπάρχει πολύ έντονη δέσμευση, πολύ εντονότερη από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, δεσμεύσεις για την απασχόληση για το, στο Plus Pack. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν πρέπει όλα αυτά να πραγματοποιηθούν τελικά, αλλά μακροπρόθεσμα λέει έχουμε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε αυτή η μακροπρόθεσμη στρατηγική αυτή τη φορά να είναι επιτυχής. Για τις ε, ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες όπως και εσείς και εγώ είμαι κάπως ε, απογοητευμένος εγώ από χαρακτήρα όμως βλέπω τα πράγματα για κάπως θετικά. Εγώ άρχισα την ε, σταδιοδρομία μου στη δεκαετία του 70 με έναν πρωθυπουργό που έλεγε ότι αποτύχαμε να έχουμε συμφωνία για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρωσεκτίας. Το 78 αυτό, ε, τώρα προχωρήσαμε. Προχωρήσαμε πολύ και υπό Βελγική Προεδρία ακόμα και με Υπουργό Οικονομικό που ορισμένοι τον γνωρίζουν καλύτερα από μένα, πετύχαμε με την ενδραμωμένη συνεργασία ένα άνοιγμα. Τώρα πρέπει να περάσουμε το τελευταίο βήμα. Είμαι σίγουρος θα περάσουν κάποιες εβδομάδες για να γίνει αυτό. Αλλά η ιδανική προεδρία, την οποία και υποστηρίζουμε, θα βρει, είμαι σίγουρος, μια λύση του προβλήματος. Υπάρχει οικονομική πτυχή υπάρχει και η κοινωνική τυχή, αν θέλετε, δηλαδή η πολιτική απασχόληση. Πρέπει να δούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να πάρουμε πολλά μέτρα. Να εργαστούμε πάνω στην ενιαία αγορά, να κοινοτοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία, να μειώσουμε τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, το επιθύμησε ο εκπρόσωπος Κομισιόδικαιος, υπάρχει το σχέδιο για τα ευρωομόλογα κλπ. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας πρέπει να γίνει στο εθνικό επίπεδο. Μπορούμε να του δώσουμε κάποια κίνητρα στις κρατικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια. Να τους πληρώσουμε ακόμα και να τους επιβάλλουν κυρώσεις όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αλλά το κύριο έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Αλλιώς πώς θα εξηγήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στη Γερμανία, την Αυστρία, τις κάτω και άλλες ζώνες της Ευρώπης του ποσοστού ανεργίας των νέων, ας πούμε, και άλλες χώρες όπου φτάνει το 50%. Τεράστιες διαφορές που οφείλονται στην πολιτική που ασχήθηκε στο παρελθόν. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε κίνητρα στις εθνικές κυβερνήσεις, στα κράτη-μέλη, για να ακολουθήσουμε τα καλά παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη το αυστριακό παράδειγμα. Δίνοντας κάποια οικονομικά κίνητρα και δίνοντας και άλλα κίνητρα. Και οι συστάσεις της Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα τα απαριθμίσω τώρα όπως το έκαναν άλλοι. Υπάρχουν λοιπόν η οικονομική πτυχή, η κοινωνική πτυχή όπως είπα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο ένωσης και τι σε επίπεδο κρατών μελών. Για τη συνθήκη, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν συγκρίνω όλα όσα είχαν λεχθεί για τη συνθήκη αυτή πριν να ολοκληρωθεί και βλέπω ότι ακούγεται τώρα, νομίζω ότι καλά εργαστήκαμε μπορέσαμε να διακανονίσουμε και μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο, κυρίως σε αυτό το κοινοβούλιο, εργαστήκαμε πάρα πολύ για να ε, σωματωθεί αυτή η διακυβερνητική συνθήκη στη, στη φιλοσοφία των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε σε μερικά, σε μερικά χρόνια η διάδοχή μας, ο δικός μου τουλάχιστον, θα μπορέσει να ενσωματώσει την συνθήκη αυτή στην συνθήκη της Ένωσης. Προσπάθησα να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή υπήρχε ο κίνδυνος που ορισμένοι πίστευαν ότι θα υπάρχει μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Πετεύχθη συμφωνία με 25, δυστυχώς όχι 27. Οκτώ που είναι εκτός Ευρωζώνης δήθηκαν αλληλέγγυοι προς εκείνους που έχουν το κοινό νόμισμα και ευρέθη μία συμφωνία ούτω ώστε εκείνοι που δεν ανοίγουν στην Ευρωζώνη αλλά επικυρώζουν τη συνθήκη να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε στιγμές κλειδιά των δυσκευτοκορυφή κορυφής της Ευρωζώνης και επίσης να έχουν ρόλο να παίξουν σε όλα τα θέματα πάνω στα οποία έχουν συμφωνήσει στη συνθήκη. Έτσι διασφαλίζαμε νομίζω κατά το δυνατόν, κατά το δυνατόν λέω, την συνοχή της Ένωσης. Και ξαναλέω, αν συγκρίνω αυτά που ελέγξαν πριν από τις διαπραγματεύσεις και αυτά που λέγουν τώρα για τη συνθήκη, βλέπω ότι πραγματικά ε, η οδός που διενήθη ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ καλή και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φανελόμπορη και για την υπομονή σας γιατί ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο που είχαμε ορίσει αλλά είναι σημαντική αυτή η συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ώρα των ερωτήσεων με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπο για εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Περιμένω λίγο να πάρουν όλες τις θέσεις τους.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 Καλώς ήρθατε, Βαρόνι.